So welcome everybody. Καλώς ήρθατε. Μας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις, παρακαλώ. Όχι από ό,τι βλέπω. ανακοινώσεις τότε του Πρόεδρου. Η πρώτη μου ανακοίνωση είναι ότι επειδή υπάρχουν πολλές συνεδριάσεις στο κτίριο σήμερα, δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε διερμηνία στα δανέζικα, τα λετονικά και τα κροατικά. Η επόμενη ανακοίνωση που έχω να σας κάνω είναι ότι έχουμε τις αποφάσεις των συντονιστών για τον ορισμό εισηγητών. Η κυρία Σιλβί Γκυγιόμ, πρώτα απ' όλα από τους σοσιαλιστές, ορίστηκε εισηγήτρια για την γνωμοδότησή μας όσον αφορά τις εκθέσεις κοντ για την απαλλαγή 2013. Η Χέλγα Στίβενς από το ECR ορίστηκε εισηγήτρια για την έκθεση σχετικά με την άδεια των χωρών μελών επικυρώσει το πρωτόκολλο 2014 για την ε, σύμβαση εξαναγκαστικής εργασίας του ILO σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν με την δικαστική συνεργασία σε ποινικά ζητήματα. Υπάρχουν αντιρρήσεις, παρατηρήσεις από αυτόν. Όχι. Οπότε έτσι φτάνουμε και στο πρώτο σημείο αυτό αυτό στην ημερήσια διάταξη που είναι η κατάσταση διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου όσον αφορά την ανάπτυξη του συστήματος e-call σε οχήματα. Παρακαλώ. Ο κύριος Άξιλ Φως. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς για το υπόβαθρο αυτού του κανονισμού. Έχουμε μια πρόταση για ένα σύστημα e-call, δηλαδή ηλεκτρονικής κλήσεως για τα νέα οχήματα, με μία παραπομπή που ε, θα σήμαινε τη σύνδεση και με το, το 112, τον αριθμό κλήσεως δηλαδή κατεπίουσες ανάγκης. Εδώ έχουμε να κάνουμε την ε, ε, κατεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικών με τον ε, ιδιώτη, στοιχεία του, στοιχεία του οχήματος, ε, ταυτότητα. Και εδώ πάλι θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι της οδηγίας του 95 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του 2002 για την ηλεκτρονική κατεργασία προσωπικών δεδομένων. Έχουμε την ΕΚΟΝ ως κύρια επιτροπή, την ΙΤΡΕ ε, και την ε, Επιτροπή των Μεταφορών όπως και την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών ως συναρμόδιες. Η δική μας Επιτροπή, ως συνδεδεμένη Επιτροπή, με το άρθρο 55, γιατί το παλαιότερο, με την παλαιότερη εκδοχή ήταν το άρθρο 50, θέλω να το διευκρίνω σε αυτό, το 55 ισχύει τώρα για μας. Είναι συνδεμένη λοιπόν η Επιτροπή, Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών τροπολογίες μπορούν να ε, υποβληθούν και χωρίς ψηφοφορίες εφόσον υπάγονται στον ε, χώρο των αρμοδίτων της Επιτροπής μας. Εδώ είχαμε μια διασυγκιστήνδα μεταξύ της Επιτροπής των ε, τη ΣΥΜΚΟ, μεταξύ Επιτροπής Ιστορικής Αγοράς δηλαδή και της δικής μας Επιτροπής για το, για το αν μπορούν οι δικές μας τροπολογίες να υποβάλλονται. Εμείς 31 Ιανουαρίου του 2014 ψηφίσαμε, στις 20, μόνο τις τροπολογίες, στις 26 εγκρίθηκε το κείμενο ολόκληρο από την Ολομέλεια και στις 8 Απριλίου, Οκτωβρίου ξεκινάει ο τριμερής διάλογος με πρώτη συνεδρίαση αύριο, Δευτέρα. Τεχνικές συνεδριάσεις έχουν γίνει μόνο μέχρι τώρα, Συμβούλιο και Επιτροπή δηλαδή. Και σκιώδεις επίσης ε, συνεδριάσεις όπως λέγονται, δηλαδή με εκπροσώπους των διαφορών πλευρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προς το παρόν διαπιστώνουμε ότι δεν είναι απλή η κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις, τη διαχείριση του θέματος από την ΕΜΚΟ αλλά και από τη δική μας την Επιτροπή, θέματα που αφορούν ε, τις αρμοδιότητες δικές μας και τη ΕΜΚΟ μπορεί να ποικίλουν αρκετά. Η κυρία Σενάλοβα από τους Ελληνικές και Δημοκράτες είναι η συγγήτρια, πρόθυμη να διαπραγματευθεί. Έχει και προτάσεις ε, στη συνεργασία με τον υποφαινόμενο. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο όμως είναι να δούμε αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον τριμερή διάλογο στο διάστημα που διαρκεί ακόμη η Ιταλική Προεδρία. Προς το παρόν έχουμε ad hoc συνεδριάσεις. Λίγες μόνο ώρες πριν από τις συνεδριάσεις βλέπουμε να μας ε, κατατίθενται τα έγγραφα θέματα δικής μας προτεραιότητας δεν βλέπουμε να έχουν υιοθετηθεί και προβληθεί. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή ιδιαίτερα φαίνεται να μην ενδιαφέρονται για προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τώρα η Επιτροπή φαίνεται να προχωράει κάπως, αλλά και το Συμβούλιο ίσως να δεχθεί κάποιες ή και αρκετές από τις δικές μας προτάσεις. Πάντως, αυτό μπορεί να οφείλεται από το γεγονός ότι και η ΙΜΚΟ έχει εντωμεταξύ πιστεί ότι είναι ευστοχιστικές μας τοποθετήσεις. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω είναι το λεγόμενο TPS, Third Part Service, η υπηρεσία δηλαδή τρίτων, προσθεφορμένη υπηρεσία από τρίτους, που ενσωματώνεται στην, ε, στο κείμενο από τρίτου ιδιώτε που μπορεί να έχουν όμω δραστηριότητα στο δημόσιο χώρο και έτσι οι συνάδελφοι τη ΣΥΜΚΟ έχοντα ε, δει τις δικές μας ε, τις δικές μας ε, παρατηρήσεις δέχονται ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεταφορά, δυνατότητα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων από το δημόσιο στο ιδιωτικό σύστημα. Το switch on, switch off, η δυνατότητα του να κλείσει κανείς το σύστημα μας έχει απασχολήσει και εδώ στην Επιτροπή μας δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε με την ΕΜΚΟ. Για το κομμάτι αυτό ε, προσπαθώ να ε, προχωρήσω σε μια έστω ε, Παναχώρησε μια ε, δεύτερη λύση, δεύτερης προτίμησης λύση που θα επέτρεπε την ακύρωση των δεδομένων, να μπορούμε να σβήνουμε τα δεδομένα, όχι το σύστημα. Αυτό είναι τώρα το θέμα συζήτησης, τουλάχιστον έχουμε ένα μόνιμο δικαίωμα διαγραφής. Πάλι πρέπει όμως να περιμένουμε τι θα πει και ο τριμερής διάλογος, θα το δούμε αύριο. Ένα άλλο ζήτημα είναι η μεταφορά των δεδομένων σε τρίτους. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι ότι αν πρόκειται να περάσει μέσα από ένα ιδιωτικό σύστημα, να απαιτείται η συνένεση του ενδιαφερομένου. Και εάν δεν, δεν έχει χορηγηθεί η συνένεση, να μην μπορεί να γίνει η μεταφορά των δεδομένων στο σύστημα από τον τρίτο ιδιώτη. Πάλι και εδώ θα ξεκαθαρίσει η εικόνα μετά τον τριμερή διάλογο. Και μια τελευταία παρατήρηση. Διελκυριστίνδα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για, το... για τις καταξουσιοδότηση και κατεφαρμογή πράξης. Εδώ ε, λέμε ότι θα πρέπει να ισχύσει η αρχή μόνο των κατεφαρμογή ε, πράξεων είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ακόμα στη συζήτηση αν θα είναι κατεφαρμογή οι εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ίσως εν τέλει μπορέσουμε να βρούμε μία λύση ώστε οι εφαρμοστικές ε, πράξεις να αφορούν μόνο τα διαδικαστικά ζητήματα, τις διατυπώσεις και η ε, κατεξουσιοδότηση να αφορούν την ουσία της εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ. Ένας θέλει να πάρει το λόγο εδώ, η Σόφη Φανχερφέλτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Άξελ για την παρουσίασή σου. Μια πρώτη παρατήρηση είναι για τη διαδικασία πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο θέλουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους τριμερείς διαλόγους όπως κάναμε μέχρι τώρα. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι δεν πρέπει να μπει στον τριμερή διάλογο, γιατί δεν πρόκειται για συζήτηση τεχνικών λεπτομεριών, αλλά πολιτικών συζητήσεων που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν χρειαζόμαστε τους τριμερείς διαλόγους, αυτοί πρέπει να περιορίζονται σε τεχνικού τύπου συζητήσεις. Και δεν είναι τεχνικό το κατά πόσο αποθηκεύονται τα προσωπικά σου δεδομένα ή όχι. Και μάλιστα δεν είναι θέμα επιλογής, είναι υποχρεωτικό τα προσωπικά σου δεδομένα, το που βρίσκεσαι, που οδηγούσες, που πήγαινες κτλ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να τα γνωρίζουν αυτά. Εγώ ήμουνα υπέρ ενός συστήματος on-off, να μπορεί κανείς δηλαδή να επιλέξει. Δεν μπορούμε να υποχρεώνουμε τον κόσμο να καταλήγει με τα δεδομένα τα αποθηκευμένα κάπου. Αναφέρατε τη δυνατότητα της ε, διαγραφής των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής, να μπορεί να γίνεται αυτό. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, τι λόγος μπορεί να υπάρχει να υποχρεώνεται ο κόσμος ή μάλλον να απαγορεύουμε στον κόσμο στο τέλος της διαδρομής να τα διαγράφει. Γιατί αν το σύστημα e-call έχει σαν μόνο λόγο ύπαρξη στην οδική ασφάλεια, τότε δεν βλέπω κανέναν απολύτως λόγο να αποθηκεύουμε δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής. Αλλιώς Υπάρχει κάτι άλλο περίεργο εδώ, πριν καν εγκριθεί αυτό το σύστημα. Και δεν θα ήθελα να εγκρίνω απολύτω τίποτα το οποίο να μην περιλαμβάνει την επιλογή αυτή. Δηλαδή, στο τέλο τη διαδρομή να μπορεί ο οδηγό να διαγράφει ό,τι δεδομένα του έχουν αποθηκευτεί. Και θέλω να ξέρω κατά πόσο υπάρχει ομοφωνία από αυτού ή όχι στον τριμερή διάλογο. Πρόεδρο, κανένα άλλο δεν θέλει το λόγο από τι βλέπω όχι, από τους σοσιαλιστές, παρακαλώ. Και μετά θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Συγγνώμη, εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Όταν λέμε ότι θα διαγράφουμε στο τέλος της διαδρομής τα δεδομένα, τότε υπάρχει καμιά ασφάλεια να ξέρουμε δηλαδή ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται ε, στην πραγματικότητα κάπου μέσα στο όχημα και όχι αλλού, γιατί δεν έχει νόημα τότε να διαγράφει κανεί κάτι το οποίο έχει αποθηκευτεί μέσα στο όχημα, αν η αποθήκευση αυτή λαμβάνει χώρα και κάπου αλλού εκτό του οχήματο. Αυτό θέλω να μου επιβεβαιώσει κάποιο, ότι η αποθήκευση γίνεται όντω σε κάποιο χώρο μέσα στο αυτοκίνητο. Πρόεδρο, αν δεν υπάρχει κανεί άλλο που θέλει το λόγο, τότε ο Αξελφός για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για τους τριμερείς διαλόγους και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την κατάσταση που έχουμε στις άλλες επιτροπές. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι ευαισθησίες τις οποίες εμείς έχουμε εδώ στην Επιτροπή μας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν υφίσταται στις ε, επίπεδο άλλων επιτροπών. Και έτσι λοιπόν η αντίληψη περί βασικών αρχών για τα προσωπικά δεδομένα, για την εξάλληψη προσωπικών δεδομένων, για την ελαχιστοποίηση, την ανανομοποίηση κτλ. των δεδομένων, από τη δική μου την εμπειρία δεν είναι επαρκής. Πρέπει δηλαδή γενικά να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Εγώ είδα ότι δεν μπορούσα να προχωρήσω στις θέσεις που θέλαμε και προχώρησα στην δεύτερη, στη δεύτερη μου επιλογή που ήταν η δυνατότητα της διαγραφής. Τεχνικά δεν ξέρω αν γίνεται. Αλλά μπορεί ίσως κάποιος να μπορεί να διαγράψει εκείνα τα δεδομένα που δεν είναι πια πλέον απαραίτητα. Σε αυτό βλέπουμε ότι επί της ουσίας υπάρχει μια συμφωνία να υπάρχει μία δυνατότητα για μόνιμη διαγραφή από τα δεδομένα, αλλά όπως είπα, αυτή η πρώτη καλή εντύπωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον τριμερή διάλογο. Αλλά φαίνεται το Συμβούλιο να είναι διατεθειμένο να το δεχθεί αυτό. Για τα ίδια τα δεδομένα τώρα. Αυτός, αυτό είναι και το σύστημα ακριβώς ε, του συστήματος του e να, να παρακρατούνται μόνο μέσα σε ένα κουτί, σε ένα box. Μόνο εφόσον χρειαστεί θα δημοσιοποιούνται, οπότε θα έχουμε τις τρεις τελευταίες θέσεις που θα κοινοποιούνται για να γνωρίζει κανείς ε, ποια είναι η κατεύθυνση που έχει λάβει ένα αυτοκίνητο από τελευταία γνωστή του θέση. Αυτό είναι κάτι άλλο, από, είναι κάτι διαφορετικό από το καθαρά υποχρεωτικό σύστημα γιατί μπορεί κανείς να έχει με ένα ιδιωτικό σύστημα δώσει τη συνένεσή του ο ιδιώτης οδηγός, επιβάτης και να πει ότι θέλει να επιτρέπει να καταγράφω τα στοιχεία του. Αυτό είναι κάτι άλλο που μπορεί να διαχειρίζεται πλέον ε, σε συμφωνία με τον κάτοχο ή τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ε, ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου, αυτοκινήτου βιομηχανία. Πάντως τα δεδομένα θα πρέπει να παραμένουν μέσα στο κουτί αυτό όπως το λέμε και μόνο εάν προκύψουν, ε, προκύψει ανάγκη, φερειπίν από ένα ατύχημα, τότε μόνο θα ε, διοχετεύονται περαιτέρω. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς και όλους τους συναδέλφους που δούλεψαν πάνω σε αυτό το θέμα. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Το θέμα αυτό είχε παραμείνει σε κρεμότητα εξαιτία του δημοψηφίσματο στην Ελβετία. Τώρα θέλω να ζητήσω από τη Ρομπέρτα Μετσόλα, που είναι η συγγήτρια εκ μέρου του ΕΛΚ, να μα εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. θέλω να συζητήσω μαζί σας για την κατάσταση πραγμάτων. Μετά την συνάντηση των σκιωδών, μάλιστα που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελβετία συμμετέχει στο σύστημα του Δουβλίνου και συμμετέχουν ενεργά μάλιστα σε αυτό. Η έχει σημαντικό ρόλο να παίξει όσον αφορά το άσυλο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι διακανονισμοί ανάμεσα στην Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτουν μία επιπλέον διάσταση. Οι ρυθμίσεις ΕΑ διακανονίζουν διάφορα πράγματα τα οποία μας συνδέουν με τις χώρες αυτές και με το Λιχνεστάν και με την Ορβηγία και ιδιαίτερα διακανονίζουν το θέμα του εύρους και της φύσης της σύνδεσης που έχουμε με την ε, Ελβετία στον τομέα του ασύλου. Πάντα πίστευα ότι η συμμετοχή της Ελβετίας στο έργο της υπηρεσίας αυτής της υποστήριξης ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Κυρίως επειδή ακριβώς ιδέονται με το σύστημα του Δουβλίνου, αλλά δεν μπορούμε τον ε, κανονισμό αυτό να το κοιτάξουμε καθαρά πολιτικά. Μετά το δημοψήφισμα στην Ελβετία υπάρχει μια νέα διάσταση στη συζήτησή μας. Θα θυμόσαστε ότι στην προηγούμενη θητεία αναρωτηθήκαμε πώς πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Πήραμε νομικές γνωμοδοτήσεις που λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχει νομικό εμπόδιο για να συναυθεί πλήρως η συμφωνία αυτή ακόμα και μετά το δημοψήφισμα. Η γνωμοδότηση όμως αυτή, η νομική αυτή γνωμοδότηση συμπεριλαμβάνει και κάποια στοιχεία τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα τελικά να μην έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των νομικών επιπτώσεων του δημοψηφίσματος που έλαβε χώρα. Επιπλέον πιστεύω ότι δεν πρέπει να βιαστούμε για να υπογράψουμε τη συμφωνία αυτή με την Ελβετία. Αν υπογράψουμε τη συμφωνία αυτή ως Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουμε ένα μήνυμα που λέει ότι συνεχίζουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα όσον αφορά την ελευθερία διακίνησης και τα θέματα μετανάστευσης με την Ελβετία. Έπειτα η Ελβετία θα διεξάγει στις 13 Νοεμβρίου και ένα δεύτερο δημοψήφισμα για παρόμοια ζητήματα. Θέση μου λοιπόν είναι να αναβάλουμε την απόφασή μας για την έκθεση αυτή σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και να περιμένουμε να έχουμε μια σαφή και λεπτομερή εικόνα των επιπτώσεων της υπογραφής μιας τέτοιας συμφωνίας με την Ελβετία. Ακριβώς επειδή έλαβε χώρα το δημοψήφισμα αυτό και θα υπάρξει και νέο. Ας αναβάλουμε λοιπόν την απόφαση γιατί έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε σε καλύτερη θέση να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις της συμφωνίας. Στο μεταξύ θα έχουμε και το αποτέλεσμα του δεύτερου δημοψηφίσματος της Ελβετίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Ματσόλα. Ένας έχει ζητήσει το λόγο. Η κυρία Βέλστρομ, εκ του Άλντε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να εκφράσω σε σας, Ρομπέρτα, τη βαθιά μου εκτίμηση για το έργο σας όσον αφορά αυτή την υπόθεση και συμφωνώ με τις απόψεις σας. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι θέση της Άλτε είναι να εγκριθεί η συμφωνία με τις διάφορες χώρες. Οπότε συμφωνώ με αυτό που λέει η Ρομπέρτα ότι πρέπει να αποφανθούμε και προτιμώ αυτό να γίνει γρήγορα παρά να καθυστερήσουμε. Βέβαια, ίσως θα ήταν όντως καλό να ξέρουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, να δούμε πώς θα ενσωματωθεί στην ελβετική νομοθεσία. Το δεύτερο αυτό δημοψήφισμα που θα λάβει χώρα σε λίγες μέρες μπορεί να περιορίσει ακόμα πιο πολύ το μεταναστευτικό κύμα προς την Ελβετία 0,2% από ό,τι φαίνεται. Οπότε συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο για μας τι σημαίνουν τα δύο αυτά δημοψηφίσματα τελικά για την Ελβετία και χρειαζόμαστε και διαβεβαιώσεις από τις ελβετικές αρχές ότι δεν θα επηρεαστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία στο βαθμό που συμμετέχει σε αυτή και η Ελβετία. Ελεύθερη κυκλοφορία για παράδειγμα που είναι και πακέτο του ασύλου ή η ρύθμιση του Δουβλίνου. Με δύο λόγια, υποστηρίζω την πρόταση της εισηγήτριας να ζητήσουμε από τη διάσκεψη των Πρόεδρων να μας δώσει άλλο ένα εξάμεινο προκειμένου να καταλήξουμε για τη συμφωνία αυτό. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό αυτό και για μας και για την Ελβετία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δύο ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο. Από τους σοσιαλιστές πρώτα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα συγγνώμη, λέει κυρία Σίπελ, εκ μέρους της συναδέρφου μου της κυρίας Σιλβί Κιγιόν που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα σας διαβάσω λοιπόν ποια είναι η δικιά της τοποθέτηση από αυτού. Πρέπει να έχουμε πιο σαφή εικόνα, όπως υπόθηκε ήδη, για τις επιπτώσεις του ελβετικού δημοψηφίσματος του Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχει λόγος και θα ήταν μάλλον καταστροφικό το να βιαστούμε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της συμφωνίας. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που μας έχουν έρθει μετά το δημοψήφισμα που μας κάνουν να θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα επόμενα βήματά μας. Πρώτον, όπως ακούστηκε ήδη, ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένη και ξεκάθαρη εικόνα των νομικών επιπτώσεων του δημοψηφίσματος αυτού όσον αφορά τους μετανάστες και ιδιαίτερα τους ετούντες άσυλο. Η έγκριση του δημοψηφίσματος αυτού αφήνει πολλά κενά και αβεβαιότητες όσον αφορά το συμβατό της τέτοια ρύθμιση με τις υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εξάλλου, έχει προγραμματιστεί στις 13 Νοεμβρίου δεύτερο δημοψήφισμα στην Ελβετία. Στόχος και περιεχόμενο της πρωτοβουλίας αυτής δεν είναι καθόλου καθισχαστικά για μας. Η νέα αυτή πρωτοβουλία θέλει να κόψει ακόμα περισσότερο τη μετανάστευση από αναπτυσσόμενες χώρες. Βάσει του ΕΚΟΠΟΠ η μετανάστευση δεν πρέπει να είναι πάνω από 0,2% του πληθυσμού κατά μέσο όρο μέσα στην επόμενη τριετία. Όπως και να έχει το πράγμα, το μήνυμα που μας φτάνει δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό. Γι' αυτό στηρίζω αυτά τα οποία ήδη υπόθηκαν, ότι δηλαδή πρέπει να αναβάλουμε την απόφαση μέχρι να έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Βερζάκ έχει ζητήσει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, υπόθηκαν ήδη τα πιο σημαντικά, συμφωνώ κι εγώ. Και ευχαριστώ την εισηγήτριά μας. Θέλω όμως να προσθέσω ότι πράγματι δεν πήγε καθόλου υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Οι συνέπειες του δημοψηφίσματος του Φεβρουαρίου δεν είναι σαφείς. Οι ελβετικές αρχές δεν μας έχουν δώσει διευκρινήσεις και θα υπάρξει και νέα δημοψήφισμα. Η μετανάστευση προς την Ελβετία δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, αλλά είναι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε πριν εγκρίνουμε την έκθεση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η συγκίτρια έχει το λόγο τώρα για να ολοκληρώσουμε. Ότι δηλαδή μάλλον αναβάλουμε την ολοκλήρωση της υπόθεσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ όλους τους κοιόδες εισηγητές που στήριξαν την θέση μου. Όσον αφορά τη διαδικασία, επειδή η προθεσμία των έξι μηνών μέσα στους οποίους η ρύθμιση αυτή θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ε, εκπνέουν, πρέπει να ζητήσουμε από τη διάσκεψη των Προέδρων να επεκτείνει την προθεσμία αυτή για άλλους έξι μήνες. Ελπίζουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα να μπορούμε να καταλήξουμε θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και πάλι από τις ελβετικές αρχές να έρθουν και να μας αναλύσουν την κατάσταση μετά από αυτό το δεύτερο δημοψήφισμα και να ζητήσουμε και από την νομική μας υπηρεσία για άλλη μια φορά γνωμοδότηση όσον αφορά το δεύτερο αυτό δημοψήφισμα. Μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά τώρα μετά το δεύτερο δημοψήφισμα από ό,τι ήταν μετά το πρώτο. Πρόεδρος, το Προεδρείο θα ακολουθήσει τις προτάσεις σας σύμφωνα με τον κανονισμό. Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν συνεργαστεί, τους ευχαριστούμε πολύ και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χρηματοδοτικά μέσα. Έχουμε μαζί μας προσκεκλημένη τη Γενική Διευθύντρια, την κυρία Μίχου, από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν το ε, πρόγραμμα εργασίας για το 2004 όσον αφορά τη χρηματοδότηση της εφαρμογής του προγράμματος δικαιοσύνη και του προγράμματος δικαιώματα, ισότητα και ηθαγένεια. Συνεπώς, το λόγο έχει η κυρία Μίχου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Μεγάλη μου χαρά σήμερα που είμαι εδώ. για πρώτη φορά, αφού υιοθετήθηκε το πολιετές πλαίσιο εργασίας, επί το οποίο δουλέψαμε, συνεργαστήκαμε μαζί σας για να βρούμε ισορροπίες ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα και ταυτόχρονα έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν και να απλοποιηθούν τα προγράμματα με τρόπο ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους και να στηρίξουν τις πολιτικές ε, δικαιοσύνης και δικαιωμάτων. Εμείς ε, είμαστε υποχρεωμένοι να ερχόμαστε και να σας αναφέρουμε την πρόοδο των προγραμμάτων αυτών Άρα λοιπόν τώρα έχουμε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας αφορά το πρόγραμμα δικαιοσύνης όπου περιλαμβάνεται η αστική αλλά και η ποινική δικαιοσύνη και το άλλο πρόγραμμα είναι αυτό που αφορά τα δικαιώματα, την ισότητα και την ηθαγένεια. Όπως γνωρίζετε, ο κανονισμό, οι κανονισμοί που θεσπίζουν αυτά τα δύο προγράμματα υιοθετήθηκαν τις τελευταίες μέρες του 2013 και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2014 για τα δύο αυτά προγράμματα, δικαιοσύνη και δικαιώματα, υιοθετήθηκαν στα τέλη Απριλίου 2014. Οι δύο αποφάσεις της Κομισιόν, οι εφαρμοστικές για τα προγράμματα αυτά, υπάρχουν στο διαδίκτυο της DG Δικαιοσύνη και περιλαμβάνεται εκεί λεπτομερής παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων επιχορήγησης και ε, διαγωνισμών που προσχεδιάζονται ε, από την ίδια αυτή διεύθυνση. Οι αποφάσεις της Κομισιόν περιλαμβάνουν επίσης μια επισκόπηση των προγραμματιζόμενων δαπανών καθώς και των ποσοστών αυτών που αποδεικνύουν ότι η κατανομή των πόρων είναι σύμφωνη με τους στόχους των συνομοθετών καθώς και με την εντολή που μας έδωσαν για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Άρα λοιπόν η ισορροπία ανάμεσα στους συγκεκριμένους στόχους διατηρείται. Τα συνολικά κονδύλια που υπάρχουν για τον προπολογισμό του 2014 για τα δύο προγράμματα ανέρχονται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τα δικαιώματα και την ισότητα έχουμε 54,2 ενώ για τη δικαιοσύνη 45,8. πάνω από το 45% θα δοθεί σε επιχορηγήσεις, ενώ το υπόλοιπο θα δοθεί σε διαγωνισμούς. Ε, θα έχουμε συνολικά 18 προτάσεις, μάλλον ε, προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που θα είναι ανοιχτέ σε επιδυνητικούς ε, υποψηφίους. 11 έχουν ήδη δημοσιευθεί, ενώ 7 θα δημοσιευθούν εντός του έτους, το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Μέσω αυτών των, ε, προτάσεων για των προσκλήσεων μάλλον για υποβολή προτάσεων, ε, στόχος είναι να προωθηθεί η πολιτική της Ένωσης για την Ιθαγένεια, ε, η πρόληψη και η καταπολέμηση ξενοφοβίας, ρατσισμού, ομοφοβίας και άλλες μορφές στήριξης της Ευρωπαϊκής Δικαστικής Κατάρτισης. Κατά την εφαρμογή του νέου προγράμματος, η Κομισιόν θέλει να ενισχύσει τη σύνδεση ανάμεσα τι πολιτικέ και τη χρηματοδότηση αυτών, καθώς και να διευκολύνει την πρόσβαση των ετούντων. Πάντοτε όμως ε, ενεργώντας μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2014 συμπεριλαμβάνει περισσότερες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τα προηγούμενα χρόνια και ότι περισσότερες εξ αυτών, και γι' αυτό ακριβώς και είναι περισσότερες, είναι πιο στοχοθετημένες σε συγκεκριμένους στόχους. Επιπλέον, οι προτεραιότητες για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ορίζονται πιο λεπτομερώς και ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις συνεχιζόμενες πολιτικές. Πολλές εξ αυτών θα πρέπει να συμβάλλουν στην ε, ε, εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στην καλύτερη ε, επιβολή των δικαιωμάτων των πολιτών επιλεγμένα προγράμματα και τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να επιδεικνύουν ισχυρή προστιθέμενη αξία, πράγμα το οποίο ήταν μέγα αίτημα που προήλθε από το Ευρωκοινοβούλιο και το έχουμε συζητήσει επί μακρόν. Ταυτόχρονος ε, στόχο έχουμε να αναζητήσουμε την ε, συνεργασία μεταξύ των ε, προγραμμάτων, το αίτημα για τα θύματα, καθώς και το πρόγραμμα των δικαιωμάτων και ο συγκεκριμένος στόχος Δάφνη και τα προγράμματα δικαιοσύνης που έχουμε συγκεκριμένο στόχο, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Όλες αυτές οι συνδυασμένες προσπάθειες γίνονται ώστε να αντιμετωπιστεί ευρύτερα ο τομέας των θυμάτων με συνεπή και ολοκληρωμένο τρόπο, καθώς και ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να επιτευχθεί μεγαλύτερος αντίκτυπος όλων των προσπαθειών. Τώρα, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η συνεργασία βασικών παραγόντων είναι μεγάλη σημασίας. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, καθώς και με βασικά ε, πανευρωπαϊκά δίκτυα και η προθεσμία εκπνέει στις 14 Νοεμβρίου και στοχεύει η πρόσκληση αυτή στην θέσπιση ε, συνεργασία και για συνεργασία σε διάφορους τομείς των διαφόρων προγραμμάτων μας. χρηματοδότηση για το 2015 για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Κατάρτισης και για το Δίκτυο ε, ε, πανευρωπαϊκών ε, συλλόγων ισότητας και αυτό προετοιμάζεται. Αλλά εμείς προσβλέπουμε στην ανάληψη δράσης για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ετούντων και όχι μόνο αυτό, αλλά για να διευκολύνουμε και τη ζωή τους σε αυτό το περίπλοκο κόσμο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που για εκείνους συχνά φαίνεται να είναι πολύ επιβαρημένος και δύσκολος. Ε, οι προσκλήσεις μας είναι ανοιχτέ σε ΜΚΟ και δημόσιους οργανισμούς και υπό ορισμένου όρους σε ιδιωτικές μορφές ε, ή πρόσωπα. Επίση, εθνικά προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν, πράγμα που επίση συζητήσαμε εδώ. Μικρά προγράμματα δεν αποκλείονται με την προπόθεση ότι αποδεικνύουν επαρκή ευρωπαϊκή προστεθέμενη αξία. Στο στόχο, με στόχο την απλοποίηση, Έχουμε έναν ενιαίο οδηγό που ισχύει για όλες τις επιχορηγήσεις αλλά και τις προσκλήσεις υποβολής ε, προτάσεων ε, και ένα μόνο ε, κανονισμό. Και αυτό έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος και εδώ το κάνουμε πιλωτικά στο Στη δικαστική κατάρτιση και αν αυτό επιτύχει θα το εφαρμόσουμε και σε άλλα προγράμματα, έτσι ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία για τους ετούντες όταν διαχειρίζονται τα προγράμματά τους, αλλά και αναφέρουν τα κόστη. Επίσης, η Κομισιόν καταβάλει πολλές προσπάθειες ώστε να διαδοθούν περισσότερο και καλύτερα οι πληροφορίες για τα νέα προγράμματα και για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Εδώ δίπλα στο, έχουμε αφήσει φυλάδια, τα οποία έχουμε εμεί εκδώσει σε όλες τις γλώσσες και είναι ενημερωτικά για τα προγράμματα τα οποία εμείς διαχειριζόμαστε. Επίσης, ε, ο ιστότοπός μας έχει αναδιοργανωθεί, ανασχεδιαστεί, ώστε να δίνει καλύτερη εικόνα για τις διάφορες ε, διαδικασίες. Έχουμε λάβει ιδέα ε, την ανταπόκριση των ετούντων που λένε ότι πραγματικά είναι πολύ πιο ικανοποιημένοι γιατί μπορούν να απλοηγηθούν ανάμεσα σε όλες αυτές τις ε, προσκλήσεις, είτε είναι αυτές που είναι ήδη ανοιχτέ, είτε αυτές που είναι για το μέλλον και μπορούν να έχουν πληροφορίες για συγκεκριμένους ε, στόχους. Επίσης, ε, ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες για τις επερχόμενες προσκλήσεις για επιβολή προτάσεων, καθώς και για τις δημοσιεύσεις με ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα. Αρκετές ενημερωτικές εκδηλώσει έχουν ήδη διοργανωθεί στα διάφορα κρατημέλη ώστε να έρθουμε σε επαφή με τους διάφορους ε, πιθανούς ε, ενδιαφερόμενους στις χώρες και να δώσουμε στοχοθετημένες πληροφορίες και καθοδήγηση για το τι γίνεται στον τομέα της δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων. Επίσης, ε, έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να αναφερόμαστε ετησίως στο Ευρωκοινοβούλιο ε, για τα επιτεύγματα των προγραμμάτων μας, αλλά όχι μόνο για τα επιτεύγματα, αλλά και για το ποια είναι τα μειονεκτήματα των προγραμμάτων αυτών κατά την εφαρμογή τους. Ε, βεβαίως, είμαστε σε πρώιμο στάδιο της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών, αλλά είμαστε μέσα στη διαδικασία προετοιμασίας της ετήσιας αυτής ε, αναφοράς. Ευχαρίστω θα σας παρουσιάσω την έκθεσή μας αυτή, την αναφορά μας και να τη συζητήσω μαζί σας, αλλά πριν να ολοκληρώσω θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε ένα ακόμα σημείο το οποίο προέκυψε μετά την αναδιοργάνωση της Κομισιόν. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Δικαιοσύνη τώρα έχει διευρυνθεί κατά κάποιο τρόπο. Λάβαμε στο, στο χαρτοφυλάκιο μας τα θέματα ε, καταναλωτή από την πρώην DG Sanko και όλα τα προγράμματα που αφορούν τους καταναλωτές, το τμήμα που αφορά τους καταναλωτές και όχι την υγεία, αυτό το έχουμε τώρα αναλάβει εμείς και οργανωτικά θα είναι μαζί μας από την 1η Ιανουαρίου, αλλά πολιτικά έχουμε ήδη ε, ξεκινήσει τη συνεργασία ε, και επίσης λάβαμε από την ε, τωρινή DG εσωτερικής αγοράς, το τμήμα που ασχολείται με το εταιρικό δίκαιο, το ενοχικό δίκαιο που τώρα καλείται ε, διακυβέρνηση εταιρική της κοινωνικής ευθύνης. Πρόκειται για ένα περίπλοκο χαρτοφυλάκιο και είμαι πεπισμένη ότι ε, με τη διαδικασία ευθυγράμμισης που έχουμε ξεκινήσει θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους ευρύς στόχους. Και φυσικά ευχαρίστως θα ξαναέρθω για να σας αναφέρω τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Μίχου. Και για την ώρα έχουμε ένα αίτημα για το λόγο. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Βερζιά και σας το δίνω κυρία Βεζιά, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω κυρίως για το θέμα του προγράμματος ε, δικαιό ε, ηθαγένεια. Οι πιστώσει στο θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ε, τρέχουσα περίοδο. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αυξάνονται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανισότητες επίσης τα πρώτα θύματα των ανισοτήτων είναι τα θύματα των διακρίσεων, τα παιδιά, οι ανάπηροι, η πλειοψηφία του πληθυσμού που είναι γυναίκες και βλέπω πολλές φορές τις ανησυχίες που εκφράζονται και στην Επιτροπή Γυναικών εδώ στο Κοινοβούλιο στην φάση ε, αναθεώρησης των διαφόρων προγραμμάτων. Επίσης, εσείς έχετε στο χαρτοφυλάκιό σας στοιχεία της προστασίας των δεδομένων, θέμα που είναι επίσης σημαντικό, το αναφέραμε και πριν από λίγο. Θεωρητικά το θέμα της ηθαγένειας είναι και αυτό τμήμα των αρμοδιοτήτων σας, ε, τουλάχιστον με βάση τα προγράμματα. Μετά δε την ε, αλλαγή της σύστασης της Κομισιόν για αυτό το θέμα ακόμα πιο πολύ διερωτώμεθα για το ποιος αναλαμβάνει αυτό το θέμα. Είδαμε να φτάνει το θέμα των δικαιωμάτων του καταναλωτή εδώ, σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, καθώς και αυτό του ενοχικού δικαίου. Η κυρία Ζουβά μας το έχει εξηγήσει και εσείς κάπως προσπαθήσατε, αλλά εγώ δεν κατανοώ πού έγκυται η λογική των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα σε όλα αυτά και πώς η κυρία Ζόλβα μαζί με τον κύριο Τίμεσμαν θα δουλέψουν για διάφορα ζητήματα, γιατί και σε δημοσιονομικό επίπεδο είναι αρκετά συγκεχημένα τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω καλύτερα ποιες είναι οι προτεραιότητες το θέμα, οι δημοσιονομικές εννοώ, ε, για το σύνολο της δικής σας διεύθυνσης. Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος, δύο ακόμα συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Πρώτα η κυρία Γκαμπριέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα επίσης να επιμείνω... Για το στο πρόβλημα, στο πρόγραμμα, Δάφνη κυρίως, απλούστευση, η οποία δεν θα πρέπει όμως να επηρεάζει την ορατότητα και τη συνοχή. Βλέπουμε έναν προϋπολογισμό 18 το 2013, 12 το 2014 εκατομμύρια, μείωση 30% και περισσότερο. Αυτά είναι τα ποσά. Και δεύτερον, έχουμε πώς μπορεί η Επιτροπή να καταπολεμήσει τις μορφές βίας κατά των παιδιών και των γυναικών, με τα ποσά αυτά, ενώ ήταν πολύ ε, ανώτερη αλλά και ανεπαρκή ταυτόχρονα η χρηματοδότηση, πρώτον και δεύτερον, αναλήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για να απλουστευθούν οι διαδικασίες οι διοικητικές, τα αιτήματα που θα επιτρέψουν έτσι και σε μικρότερε με κυβερνητικές οργανώσεις να προτείνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Δάφνη. Πώ δηλαδή μπορεί να βελτιωθεί και η ορατότητα μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και να διαφυλαχθεί το ίδιο. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αποτελεσματικότητα και είναι και πολύ δημοφιλέ. Ευχαριστώ. Κυρία Στίβενς. πει αξιότιμοι συνάδελφοι. Έχω μια ερώτηση καταρχάς. Θέλω να ευχαριστήσω για τις εξηγήσεις που μας δίνετε για το πολύ ενδιαφέρον αυτό πρόγραμμα. Έχω μια ερώτηση. Προτείνεται ένα συμπληρωματικό προπολογισμό για κάποιου οργανώσει ή οργανισμού που εργάζονται με άτομα με αναπηρία δεδομένου ότι αυτό συνεπάγεται επιπλέον κόστος. Έχουμε κοφαλάλους, έχουμε κοφούς με δυσκολία γραφής και που χρειάζονται κάποιον που μπορεί να τους βοηθήσει ή έχουν ε, διανοητικούς περιορισμούς και χρειάζονται κάποιου άλλου τύπου πλαισίωση. Εγώ πάντως αναφέρομαι στο, ε, ε, στην επιπλέον επιβάρυνση που σχετίζεται με την αναπηρία, γιατί οι λοιπές ομάδες δεν, δεν επιβαρύνονται. ασφαλώς και θα πρέπει τα άτομα αυτά να μπορούν να, να έχουν πρόσβαση καλύτερα στα προγράμματα αυτά. Μια πιο δημοκρατική κοινωνία σημαίνει και καλύτερη ε, προστασία βεβαίω των προσωπικών του δεδομένων και όλα αυτά. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν ειδικέ διατάξει για τα άτομα με αναπηρίε ω ομάδα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά. Γιατί όπως είπαμε, πολλές φορές επιβαίνονται με πλέον δαπάνη και έτσι διαπιστώνουμε, στο παρελθόν τουλάχιστον, ότι ε, απορρίπτονται οι προτάσεις τους λόγω κόστους. Ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούνται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικές ερωτήσεις το ετήσιο πρόγραμμα. Παρακαλώ την κυρία Μίχου λοιπόν να μας απαντήσει για ένα τελικό γύρο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος καταγράφονται αναστόχως το νηστότοπο μας. Δίνουν δε συγκεκριμένα στοιχεία για το τι ποσά προβλέπονται για το κάθε στόχο. Θέλω όμως και να διευκρινίσω ότι εάν, επί παραδείγματα, εξετάζουμε το Δάφνε ή άλλα προγράμματα, Πρέπει να κοιτάξουμε και τα δύο προγράμματα. Αυτή τη φορά και όπως είπα και στα εισαγωγικά μου σχόλια, δεν εξετάζουμε μόνο όπως συνέβαινε πριν, μόνο το Δάφνη με τίτλο Δάφνη και δίπλα το ποσό που αντιστοιχεί. Τώρα μιλάμε για το Δάφνη και πρόσβαση στο πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη. Συνδυαζόμενα λοιπόν αυτά τα δύο προγράμματα μας δίνουν ένα ποσό υψηλότερο από αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν έρθουν τα στοιχεία εκ των υστέρων με την έκθεση που θα υποβάλουμε το 2015 θα τα δείτε. Οι διάφοροι τομείς που αναφέρατε τώρα. Όλοι αυτοί οι τομείς έχουν καλυφθεί ή θα καλυφθούν στα προγράμματα που δημοσιεύουμε ή που θα δημοσιεύσουμε. Αυτό που θέλω να επισημάνω πάντως είναι το εξή ότι εμείς δημοσιεύουμε τον ιστότοπο, διαθέτουμε τις πληροφορίες στον ε, καθένα, ε, μεταβαίνουμε στα κράτη-μέλη για να τα ενημερώνουμε για τα προγράμματα. Είστε και εσείς εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις, τους διάφορους φορείς να συμμετέχουν και πραγματικά ζητώ την υποστήριξή σας και σας καλώ να μας ε, επισημαίνετε ή να ε, βοηθάτε με τη συμμετοχή σας σε συγκεκριμένους τομείς. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να πάω σε μια περιοχή και να κάνω μια αναγγελία λέγοντα πρέπει να συμμετάσχετε, να κάνετε αίτηση. Εμεί προσπαθούμε να κάνουμε στο δυνατόν πιο γνωστό το πρόγραμμα, να διαδώσουμε την πληροφορία. Πιστεύω ότι αν δουλέψουμε όλοι μαζί για να διαδοθούν τα αποτελέσματα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε και πιλωτικά προγράμματα, τα οποία προτείνετε εσείς. Και προσπαθούμε να συνδυάσουμε αυτά που μας έχετε προτείνει μέσα στο πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα ήθελα, παραδείγματι, να αναφερθώ στην κατάρτιση με τον κύριο Μπερλιγκουέρ και άλλους ε, βουλευτές ή στο πρόγραμμα για την ε, γλώσσα για κοφαλάλους που μας βοηθήσατε με τον τρόπο σας να υλοποιήσουμε τα προγράμματα τα οποία προσπαθούμε να τα έχουμε στο δυνατόν πιο απλά, πιο αποτελεσματικά και χρήσιμα για τον ωφελούμενο, τον δικαιούχο, αλλά και για μας. Γιατί, γιατί είμαστε 5-6 διαφορετικές μονάδες που διαχειρίζονται τα οικονομικά. Τώρα τα έχουμε διοχετεύσει σε μία μονάδα υπό μία διεύθυνση προκειμένου να υπάρχει ο ενιαίος οδηγός για τον κάθε ε, τούντα, ε, ίδιες προταγραφές και προϋποθέσεις κτλ. Και χωρίς να λέω ότι είμαστε τέλειοι και δεν θέλουμε να μάθουμε ε, τίποτε καινούριο, Πρέπει να επισημάνω ότι βρισκόμαστε στην αρχή του δημοσιονομικού έτους. Προσπαθούμε λοιπόν να προσαρμόσουμε τις ελλείψεις σε σχέση με αυτά που θα δούμε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους. Τώρα να τελειώσω με την ηθαγένεια. Ξέρω ότι επικρατεί μια σύγχυση για το τι κάνει ποιος με στην Επιτροπή. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ανέλαβε το πρόγραμμα Ιθαγένεια. Η δική μας η Γενική Διεύθυνση συνεχίζει να κάνει αυτό που έκανε και πριν, δηλαδή δικαιώματα των πολιτών ή συνδεόμενα με την ηθαγένεια. Αυτό ήταν και το πράγμα που είχαμε συζητήσει μαζί σας. Θα προσπαθήσουμε τώρα, μαζί με τους συναδέλφους τη Γενικής Διευθύνσης των Εσωτερικών, να εξετάσουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ή να βάλουμε, να σπρώξουμε προ την ίδια Αλλά αυτό που άλλαξε ήταν η DigiCom και το πρόγραμμα, η Γενική Διεύθυνση δηλαδή Επικοινωνία και παραμένει το πρόγραμμα υπό τον κύριο Αβραμόπουλο με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μας μιλήσετε, να μας εξηγήσετε το πρόγραμμα. Η, συνεχή, η Επιτροπή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να ελέγχει βέβαια. Ευχαριστώ. Στο επόμενο θέμα. Πάλι ευρωπαϊκό πρόγραμμα για χρηματοδοτικά μέσα, σχετικό με την όλο αυτή τη φορά. Έχουμε τον Γιώχαν Κόου, επικεφαλής της ομάδας της Όλαφ D5. Καλώς ήρθατε. Ο οποίος θα παρουσιάσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2014 για την ανταλλαγή, σύνδρομη, κατάρτιση σε σχέση με την προστασία του ευρώ κατά της ε, παραποίησης, το πρόγραμμα Περικλής 2020. Κύριε Κόου, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, εξαιρετική ευκαιρία όντω ε, που προσφέρετε στην Επιτροπή να έρθουμε ενώπιον τη Επιτροπή σα και να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα Περικλής 2020 και το ετήσιο πρόγραμμα εργασία. Θέλω να σας προσφέρω κάποιες πληροφορίες σαν υπόβαθρο και να εξηγήσω και κάποιες ιδιαιτερότητες του προγράμματος ε, εργασίας για το 2014 και θα κοιτάξω και προς το προς. Το πρόγραμμα λοιπόν Περικλής είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής σύνδρομης και κατάρτισης για την προστασία του ευρωκατά της ε, παραποίησης. Ιδρύθηκε, θεσπίστηκε με μια απόφαση του Συμβουλίου του 2001 και με απόφαση που κάλυπτε την περίοδο 2002-2005 και έχει εντωμεταξύ παραταθεί η λειτουργία του από το 2006 στο 2013 με άλλες αντίστοιχε αποφάσεις. Έως τις 11 λοιπόν Μαρτίου εφέτος υιοθετήθηκε το πρόγραμμα Περικλής 2020 για την προγραμματική περίοδο 14-20 στο πλαίσιο του πολιτισμού συνομικού πλαισίου. το βασικό νομοθέτημα έτεθε σε εφαρμογή στις 6 Απριλίου του 2014. Η υλοποίηση του κανονισμού υπό αριθμών 3031 αφορά μόνο τα κράτη της Ευρωζώνης. Συμπλήρωμά του δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή, διότι εκκρεμεί η κύρωσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το προηγούμενο πρόγραμμα Περικλής αφιέρων 7 δις για την περίοδο 2007-2013. Εφαρμόστηκε κατά τρόπο επιτυχή μπορούμε να πούμε με 113 έργα που υλοποιήθηκαν, 72 έργα που παρήχθησαν από τις αρμόδιες αρχές των αρμοδίων ε, αρχών, κυρίως ε, αστρομικές αρχές, αλλά και εθνικές ε, κρατικές τράπεζες αλλά και εθνικά νομισματοκοπία και ένα 30% περίπου ήταν η παραγωγή της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Όλαφ. Στην περίοδο 2007-2013 είχαμε 4.320 εμπειρογνώμονες που συμμετέσχουν σε προγράμματα προερχόμενοι από 83 διαφορετικές χώρες και η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση έγινε μια φορά το 2013 και μια φορά το 2014. Σας κοινοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Είχε αποδειχθεί ότι το προηγούμενο πρόγραμμα δεν ήταν αποτελεσματικό. Συγγνώμη, απειδείχθη ότι ήταν αποτελεσματικό και έφερνε ουσιαστικά αποτελέσματα παρότι ήταν το πιο μικρό σε προπολογισμό πρόγραμμα. Για το 2020 λοιπόν και τον κανονισμό 3031 του 2014 μπορούμε να πούμε ότι έχει προσφέρει 7,3 εκατομμύρια ευρώ για την ευθαετία σε τωρινές τιμές ευρώ και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020. Στόχος του προγράμματος είναι να αποτρέψει και να καταπολεμήσει την παραποίηση και την ε, απάτη που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την βιωσιμότητα των ε, δημοσιονομικών μας. Το πρόγραμμα είναι εξυγχρονισμένο, απλουστευμένο, ιδιαίτερα σε σχέση με, τα επιλέξη, με τις επιλέξιμες δαπάνες και τους εθνικούς φορείς που μπορεί να ορίσει ο Ευρωπαίος Νομοθέτης. Ο κανονισμός ορίζει επίσης ενισχυμένες διατάξεις παρακολούθηση επιπτίας αξιολόγησης υποβολής εκθέσεων από τα στοιχεία που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοιχεία που αφορούν τους Δικαιούχου βέβαια. Αυτή η λογοδοσία σημαίνει για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τακτικότερη και πιο πιστή ε, ενημέρωση για την εφαρμογή του προγράμματος Περικλής το οποίο επίσης προβλέπει διάταξη για κατεξουσιοδότηση πράξη από τι Ευρωπαϊκέ Επιτροπέ. Πώ εφαρμόζεται αυτό. Με βάση το βασικό κείμενο του κανονισμού, τη βασική πράξη, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα υιοθέτησε το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα η Επιτροπή το Μάιο του 2014. Υιοθετείται λοιπόν το πρόγραμμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υλοποιεί επί τη βάση του κανονισμού μέσω επιδοτήσεων, ενισχύσεων, δωρεών, στοχεύοντας ιδιαίτερα περιφέρειες που διαπροσωπεύουν κίνδυνο σε σχέση με την παραποίηση ή την παραχάραξη του νομίσματος. προβλέπονται αυτές οι λεπτομέρειες, συνεργαζόμαστε με τους εμπειρογνώμονες μέσω ε, σεμιναρίων, διασκέψεων, εργαστηρίων κατάρτισης, πρακτικής ανταλλαγής, ε, πρακτικής εξάσκησης ανταλλαγών, εμπειρογνωμόνων και λοιπόν δραστηριοτήτων που διεξάγονται τόσο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής, αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2014 καλύπτει 925 περίπου χιλιάδες ευρώ και στηρίζεται στη στρατηγική περικλής. Η στρατηγική περικλής είναι ένα, ένα έγγραφο το οποίο έχουμε καταρτήσει συνεργασία με τους ειδικού ε, σε θέματα παραχάραξης από τα κράτη-μέλη, από τις αστυνομικές αρχές και από τις τράπεζες, αλλά βέβαια και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη Europol και με τους οποίους ορίσαμε και συστήσαμε και ορίσαμε τις ε, προτεραιότητες του Περικλή. Πάντοτε ενήμεροι για το ποιες είναι οι τελευταίες και πιο πρόσφατες απειλές σε σχέση με την ε, παραχάραξη ή απομιμής του νομίσματος μέσα στην Ένωση εκτός αυτής και πάντα σε σχέση με το ευρώ. Οι προτεραιότητες. που καταγράφονται με το πρόγραμμα 2014 είναι αυτές στις οποίες εντοπίστηκαν κύριες ανάγκες, δηλαδή εκεί όπου η παραχάραξη θα μπορούσε να αποτελέσει μια πραγματική ε, απειλή σε ένα συγκεκριμένο κράτος. Ιδιαίτερα εστιαζόμαστε στην ε, νοτιοανατολική περιοχή των Βαλκανίων ε, και την Τουρκία, αλλά γενικότερα κοιτάμε που υπάρχει ιδιαίτερο κίνδυνο σε σχέση με την παραχάραξη του ευρώ. Η περιοχή του Μαγκρέβ επίση ε, είναι στους στόχους μας. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές της Γαλλίας και της Ιταλίας ώστε να μελετήσουμε πιο προσεκτικά αυτή την περιοχή όπου έχουμε ζήτημα παραγωγής, παραχάραξης χαρτονομίσματος και νομίσματος ή κυβδηλίας. Ε, τελευταία, ε, επίσης, ε, ασχολούμαστε και με τη Λατινική Αμερική, αφού η Κολομβία αποτελεί ένα σημείο κρίσιμο, ένα χώρο κρίσιμο για την παραχάραξη, spot όπως τα λέγαμε, όχι μόνο του ευρώ αλλά και του δολαρίου. Άλλωστε αυτή η παραχάραξη είναι μέρος μιας ε, πολύ ευρύτερης εγκληματικής δραστηριότητας που έχει να κάνει και με νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων και με ελαθρεμπόριο κοκαίνης από την περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν μας απασχολούν και τα θέματα της Κολομβίας. Υπάρχουν διάφοροι τομείς όπου κάνουμε κατάρτιση στις εθνικές αρχές και συνεργαζόμαστε με τις αρχές ε, καταστολής. Για το 2014 τώρα και την εφαρμογή του προγράμματος, αφού ήδη έχει περάσει το μισό έτος από την ε, θέση στη λειτουργία ή την ε, υλοποίηση, έχουμε δημοσιεύσει μια πρώτη πρόταση υποβολής ενδιαφέροντος για 640 εκατομμύρια ευρώ για χορηγίες με την εκπνοή της προθεσμίας είχαμε τέσσερις αιτήσει, εκ των οποίων στις τρεις δόθηκαν χορηγίες. Έχουμε τις εθνικές αρχές, ήταν σχέση με την Κολομβία, όπου γίνεται η κατάρτιση και στις, ε, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κτλ. Υπάρχει ένα ε, μια χορηγία από την γαλλική Πολυζουτισιέχ, τη δικαστική αστυνομία, που καλύπτει όχι μόνο το ιστορικό της Γαλλίας αλλά και εκτός Γαλλίας δραστηριότητες παραχάριξης και στοχεύει στην αποδιάρθρωση των δικτύων διάθεσης μέσα στη Γαλλία και επίσης έχουμε ένα ε, έργο ιταλικό που προτάθηκε με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικού σε σχέση με το Μαγκρέπ, με τις χώρες εταίρους, αλλά και με εκπροσώπους της Ισπανίας και της Γαλλίας. Άλλο τμήμα του προπολογισμού δαπανάται για συγκεκριμένες δράσεις και με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με έναν ε, υπεργολάβο, ο οποίος αναλαμβάνει την οργάνωση σεμιναρίων και εργαστήριων ε, ε, σε συνεργασία πάντα και στη συμμετοχή των ε, τεχνικών εμπειρογνωμόνων ειδικών και έχουμε τη φιλοδοξία αυτές οι πράξεις εξουσιοδοτημένες όπως θα τις λέγαμε να συνεχιστούν. Έχουμε και ένα ειδικό εργαστήρι, workshop για τις τουρκικές αρχές, αφού η Τουρκία ως χώρα εκπροσωπεί ένα κάποιο κίνδυνο και παραχάραξη του ευρώ, είναι και πολύ μεγάλη χώρα και υποψήφια χώρα. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει μαζί με τους εμπειρογνώμονες και βάσει αξιολογήσεως κινδύνου να ξεκινήσουμε αυτή ε, την συνεργασία από το 2015 μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Europol έχουμε και την τρίτη διεθνή διάσκεψη για την προστασία του ευρώ που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Φραγκφούρτη, στα νέα κεντρικά γραφή της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να καλυφθούν όλα τα θέματα παραχάραξης και κυβδηλίας του ευρώ. Και επίσης τελευταίο θέλουμε να δώσουμε ειδική κατάρτιση για τους ε, ε, για την περιοχή του Κάλι στην Κολομβία, εκεί δηλαδή που διαγνώσκονται οι υψηλότεροι κίνδυνοι παραχάραξη και κυδηλία. Ε, πώς γνωρίζετε βέβαια, για να ολοκληρώνω, η προστασία του ευρώ με, το πρόγραμμα Περικλές προχωράει με απόφαση του Προέδρου ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Όλαφ περνάει στα χέρια της DG ECFIN, από όλες δηλαδή τις υπηρεσίες που ήταν αρμόδια ή μόνο αρμόδια η DG ECFIN, από τις αρχές Νοεμβρίου με τον Επίτροπο Μοσκοβισή και τον κύριο Μάρκο Πούτ, που νέος, ο τωρινός διευθυντής. Επομένως, όπως είπα, μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες από την Όλαφ στη DG ECFIN για τα θέματα της χάραξης πολιτικής. Από τις 5 Νοεμβρίου η οργάνωση και το οργανόγραμμα ισχύει από 1η Πρώτη του 2015, όπως ξέρετε. Ο κ. Μασκοφίση λοιπόν είναι τώρα υπεύθυνο και για την προστασία από την παραχάραξη και την κυβδηλία του Ευρω... Ε, και το πρόγραμμα Περικλής. Συνεχίζουμε την επιτήρηση και την ε, παρακολούθηση του προγράμματος 2014 εμείς, όπως Κάθε φορέας ε, διαβιβάζουμε σε εσάς έκθεση λεπτομερή για την εφαρμογή στα αρχές του 2015 την εφαρμογή του 2014 όπως και το άρθρο 13 και συνεχίζουμε τις συζητήσεις στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την πλαστογραφία παραχάραξη και βέβαια συνεχίζουμε να πιέζουμε και να καλούμε τον Ηνωμένο Βασίλειο να κυρώσει την παράταση της λειτουργίας του κανονισμού για την περίοδο αυτή έως το 2020. Τα κράτη που έλαβαν μέρος ε, μέχρι τώρα έχουν επιδείξει πολύ καλές επιδόσεις και θέλουμε με την ε, κύρωση αυτή από το να προχωρήσει σε ολοκλήρωση το πρόγραμμα όσο το δυνατόν ταχύτερα. Ευχαριστούμε. Ήταν αρκετά πλήρες. Εγώ τουλάχιστον δεν είδα να θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για τη στήριξη του προγράμματος αυτού και την εφαρμογή του. Θα παρακολουθήσουμε από κοντά τη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Χρηματοδοτικού προγράμματος για δράση της Ένωσης τα πλαίσια του ασύλου εσωτερικής ασφάλειας, εξωτερικά σύνορα και θεωρήσεις, αλλά και όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία. Φιλοξενούμενος μας είναι ο κύριος Σίγκαν, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Home Εσωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε, κυρία Τσίγκαν, και σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές της Επιτροπής ΛΥΜΕ. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω και να σας μιλήσω για τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκατε. Αναφερθήκατε στο ετήσιο πρόγραμμα 2014 για την χρηματοδότηση της δράσης της Ένωσης και της έκτακτης βοήθειας. Όπως ξέρετε, υπάρχουν τα κονδύλια για τα εθνικά προγράμματα. Θα θυμόσαστε ε, τα δύο που είχαμε για να στηρίξουμε τις πολιτικές μας για την περίοδο 2014-2020 για τη μετανάστευση και την εσωτερική ασφάλεια, ότι είχαν δηλαδή σχεδιαστεί αυτά προκειμένου να έχουν στα στόχο τη σωστή πολιτική, αλλά από την άλλη μεριά να είναι ευέλικτα και πιο απλοποιημένα. Σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να επικεντρώνονται πολύ καλύτερα στα αποτελέσματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο αυτά κονδύλια μπορούμε να τα διαχειριστούμε με δύο τρόπους. Μέσω εθνικών προγραμμάτων, με μεταφορές και με μεταφορές στις χώρες μέλη. Και μετά οι αρμόδιες αρχές των χωρών μελών τα διαχειρίζονται. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να έχουν προηγουμένως υποβληθεί τα εθνικά προγράμματα. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και αποκεντρωμένη διαχείριση, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη η οποία αποφασίζει για το πού θα πάνε τα χρήματα και τότε η διαχείριση γίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των ετησίων προγραμμάτων εργασίας. Κάτι που είναι σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε ότι στη νέα αρχιτεκτονική των κονδυλίων Home τα ετήσια προγράμματα εργασίας παρά τη φύση τους που κανονικά είναι ετήσια σχεδιάζονται με μια πολυετή προοπτική δηλαδή τα προγράμματα που σχεδιάζονται για το 2014 έχουν μία σχέση με τα προγράμματα δράσης τα προηγούμενα και τα επόμενα. Η έγκριση του ετησίου προγράμματος εργασίας για το 2014 ήταν μεγάλη πρόκληση για μας επειδή οι βασικές ρυθμίσεις άργησαν να υιοθετηθούν επειδή είχαμε τις ε, δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις θα θυμόσαστε. παρόλα αυτά εγκρίναμε τρία ετήσια προγράμματα για την αστυνομία ISF που εγκρίθηκε στις αρχές του Αυγούστου με 100 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Αυτό έθεσε το πλαίσιο και άνοιξε το δρόμο για να αρχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εσωτερικές υποθέσεις. Έτσι, μετά από διαβούλευση με τις χώρες μέλη, ίσως να θυμόσαστε ότι όταν συζητήσατε την κατάσταση πραγμάτων των εθνικών προγραμμάτων, ένα από τα ενδιαφέροντα ε, σημεία ενημέρωσης ήταν ότι για πρώτη φορά χρησιμοποίησαμε αυτό που για πρώτη φορά φτιάχτηκε, που είναι ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συναντιούνται και να συζητούν διάφορες πολιετής προτεραιότητες για τα επόμενα 7 χρόνια. Αυτό έγινε στα πλαίσια της προετοιμασίας για τα εθνικά προγράμματα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο μας. Όταν όμως έχουμε τις συναντήσεις αυτές, χρησιμοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να συζητήσουμε με τις χώρες μέλη και να δούμε τι είδους προγράμματα θα μπορούσαν να τα ενδιαφέρουν και σε ποια από αυτά θα υπήρχε μια ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκαν οι προτεραιότητες βάσει των ε, πολιτικών προτεραιοτήτων εσωτερικών υποθέσεων αλλά και ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν. Το δεύτερο στοιχείο τώρα που θέλω να σας εξηγήσω είναι ποιο ήταν οι κύριες πτυχές που λάβαμε εμείς υπόψη μας για την προετοιμασία των ετησίων προγραμμάτων εργασίας. Για μας το πρώτο στοιχείο που λαμβάνουμε υπόψη είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διασυνοριακές δράσεις και με και που να ανταποκρίνονται σε γενικότερες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Το άλλο που συζητήσαμε είναι η συμπληρωματικότητα με τα εθνικά προγράμματα, τα μελλοντικά εθνικά προγράμματα. Και εδώ πανέρχομαι στον μηχανισμό που χρησιμοποιούμε αυτό, όταν έχουμε διάλογο και συζητάμε για τα μελλοντικά προγράμματα δράση. συγκεντρώνουμε όπως καταλαβαίνετε πληροφορίες έτσι ώστε αργότερα να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την συμπληρωματικότητα με τις εθνικές δράσεις. Ένα άλλο σημαντικό και νέο στοιχείο είναι οι διασυνοριακές πρωτοβουλίες οργανισμών, προκειμένου στην πράξη να υπάρχει συνεργασία. Πολύ σημαντικό στοιχείο στην εφαρμογή των πολιτικών μας. Ένα άλλο στοιχείο είναι η εξωτερική διάσταση και η συμπληρωματικότητα με άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, διαφορετικά ταμεία, κοινωνικό ταμείο, περιφερειακό ταμείο και άλλα μέσα εξωτερικής δράσης. Άρα και εδώ μπορούμε να εξετάσουμε τη συμπληρωματικότητα για να αποφεύγουμε επικαλύψεις ή κενά ενδεχομένως. Τέλος, ένα άλλο στοιχείο είναι το θέμα της έκτακτης ανάγκης και αυτό αποτελεί μέρος των ετησίων προγραμμάτων εργασίας μας και θα επανέλθω αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για τα τρία ε, κείμενα. Μπορείτε να τα βρείτε. Εγώ μπορώ επίση να σας τα στείλω αν θέλετε, αλλά θα σας δώσω κάποια παραδείγματα με τα ποσά. Έτσι είσαστε καλύτερα σε θέση να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται για το άσυλο, μετανάστευση και ένταξη για το 2014 προβλέπουμε 37,4 εκατομμύρια, από τα οποία 25 πηγαίνουν σε έκτακτη ανάγκη και τα υπόλοιπα για διάφορες δράσεις. Τα παραδείγματά μου είναι προγράμματα και δράσεις. Ένα πολύ ενδιαφέρον είναι για τον εντοπισμό και τις πρόθεσεις των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του ασύλου. Εντοπίζουμε δηλαδή τις ειδικέ ανάγκες παιδιών και γυναικών κύρια, πώς θα έχουν πρόσβαση στις νομικές διαδικασίες και την ενημέρωση δωρεάν και πώς εντάσσονται οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Ένα άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα για το μέλλον των εκστρατιών ενημέρωσης. Εκστρατείες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αποφεύγονται κίνδυνοι σε βάρος ε, παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες και δεν έχω παραδείγματα και επευκαιρία σας λέω ότι συνεργαζόμαστε για αυτές τις δράσεις και με οργανώσεις όπως είναι των Ηνωμένων Εθνών ή άλλοι. Με τις υπηρεσίες ε, του ΟΗΕ, δηλαδή που ασχολούνται με την Αιθιοπία και το Σουδάν, μεταξύ άλλων. Εδώ λοιπόν κοιτάμε πώς έχει γίνει η εφαρμογή και τι δράσεις θα έπρεπε να εφαρμοστούν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δοθεί συνέχεια σε αποφάσεις που ελήφθησαν από την Task Force για την Μεσόγειο. Ένα παράδειγμα λοιπόν για την ασφάλεια και την ένταξη των ε, μεταναστών θυμάτων από την εμπορία το 2004 αποφασίσαμε να ασχοληθούμε περισσότερο με την Αλβανία, το Μαρόκο και την Ουκρανία. Και εδώ θα αναφέρω το άμυφ. Είναι ένα παράδειγμα διασυνοριακή συνεργασία, Είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που είναι η διευκόλυνση κινητικότητας και εταιρικής σχέσης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα του 2014 όχι μόνο για την μετανάστευση και την ένταξη, αλλά και για την εσωτερική ασφάλεια. Είναι ένα καινοτόμο εργαλείο, όπως σας είπα, που στηρίζουν όλοι, γιατί θέλουμε να είναι ευέλικτο και να βοηθάει χώρες που συνεργάζονται μαζί μας όσον αφορά την εταιρική σχέση κινητικότητας. Και εδώ πάλι πρόκειται για την εφαρμογή που οδηγεί σε βελτίωση της συνεργασίας. Όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις, έχουμε 15,7 εκατομμύρια, 8,9 είναι για δράσεις και τα υπόλοιπα για εκτακτή βοήθεια. Και να σας δώσω εδώ κάποια παραδείγματα δράσεων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο αυτό πρόγραμμα εργασίας. Αυτά έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση του Σέγγεν, με τη συνεργασία Eurosur, συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών, στήριξη τεχνικών ικανοτήτων χωρών μελών προκειμένου να εντοπίζουν μικρά σκάφη στη θάλασσα. Είναι εδώ και η περιφερειακή συνεργασία, η διαχείριση συνόρων, σε συνεργασία χωρών μελών με τρίτες χώρες. Πολύ συχνά επίσης πρόκειται για προγράμματα περιφερειακά κατάρτισης. Έχουμε εδώ και την ενίσχυση τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Πολύ βασικό. Γιατί μερικές φορές έχουμε να κάνουμε με πολύ περίπλοκα ζητήματα διαχείρισης ε, συνόρων. Όσον αφορά τώρα την αστυνομική συνεργασία στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, εδώ έχουμε 49,5 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 50. Δεν υπάρχει εδώ εκτακτή βοήθεια. Παραδείγματα είναι η πρόθεση της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου, την αντιμετώπιση της διαφθοράς, των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, των σεξουαλικών εγκλημάτων, στήριξη επίσης ευρωπαϊκών δικτύων, που το γνωρίζετε όπως είναι το Atlas ή η συμβουλευτική ομάδα. Υπάρχουν και δραστηριότητες για τον αστυνομικό κύκλο 14 με 17 και άλλα παραδείγματα για την αντιμετώπιση εμπορίας ατόμων, επικοινωνίας και ευρωβαρόμετρο όσον αφορά το κυβερνοχώρο. Αλλά υπάρχει εδώ και η συνεργασία στον τομέα της έκτακτης ανάγκης. Θα έχετε διαπιστώσει ότι είπα πως το πρόγραμμα εγκρίθηκε αρχές Αυγούστου. Άρα οι δράσεις προβλέπονται για τους τελευταίους μήνες. Οπότε τώρα ε, δημοσιεύουμε ε, προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Φροντίζουμε όλα αυτά τα προγράμματα να ξεκινήσουν και είναι σε διαφορετικά στάδια εφαρμογής το καθένα. Εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και θα τελειώσω με το εξής για την έκτακτη βοήθεια. Αποτελεί μέρος των ετησίων προγραμμάτων εργασίας. Είναι ενδιαφέρον να τον διαφέρουμε εδώ γιατί αν συγκρίνουμε τι γινόταν στον προηγούμενο μηχανισμό, το μηχανισμό εκτακτής βοήθειας, υπάρχουν αλλαγές. Και οι αλλαγές αυτές έχουν ως στόχο να γίνει πιο ευκολόχρηστο το μέσο αυτό για να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε απρόοπτες καταστάσεις μεταναστευτικών πιέσεων που έχουν να κάνουν και με την εσωτερική ασφάλεια. Το πρώτο βασικό είναι ότι η αρρωγή αυτή μπορεί να είναι 100% του, της επιλεγμένης δαπάνης. Και το δεύτερο είναι για να διευκολυνθεί και να απλοποιηθεί η διαδικασία. Είναι λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη δεν χρειάζεται να αλλάξουν τα προγράμματά τους για να πάρουν αυτή την έκτακτη βοήθεια. Αποτελεί μέρος του ετησίου προγράμματος εργασίας. Χρειάζονται μετά κάποια βήματα βέβαια, αλλά η όλη διαδικασία είναι πιο εύκολη. Δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Η αναθεώρηση των εθνικών προγραμμάτων ήταν κάτι πολύ βαρύ στη διαδικασία. Επεκτείνεται επίσης και το εύρος εφαρμογής. Τώρα έχουμε και την εξωτερική διάσταση, την δυνατότητα έκτακτης αρρωγής και υπάρχει το θέμα της αστυνομικής συνεργασίας που προβλέπεται για το 2015 και μετά. Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι πριν την περίοδο εφαρμογής είχαμε έξι μήνες. Ενώ τώρα μιλάμε για 12 μήνες ήδη από το 2014. Άρα έχουν περισσότερο χρόνο οι χώρες μέλη για να θέσουν σε εφαρμογή τα διάφορα μέτρα. Η δαπάνη στήριξη και η αίτηση για αρρωγή είναι πράγματα που επίσης υπάρχουν και μπορεί να είναι χρηματοδοτικά μέσα απευθεία από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Το ποσό λοιπόν, αν ρωτάτε γιατί έχουμε αυτά τα ποσά και όχι άλλα για το 2014, αποφασίστηκαν βάσει ανάλυσης αναγκών και εμπειρίας που έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια. Το 2014 είναι βέβαια λίγο ιδιαίτερη χρονιά επειδή υπήρξε η έγκριση πολύ αργά. για το ΑΕΣΕΦ έκτακτη ανάγκη είναι 6,8 και ήρθαν σε επαφή μαζί μας μέχρι τώρα πολλές χώρες με η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος. Έχουμε μία επίσημη αίτηση από την Κύπρο την οποία εξετάζουμε σήμερα. Θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες μας λαμβάνοντας υπόψη το κριτήρια του συμβατού, της ποιότητας της πρότασης, των ε, οικονομικών επιπτώσεων κλπ. Μετά την αξιολόγηση αυτή μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Όσον αφορά τώρα το Ταμείο για το Άσυλο Μετανάστευση και Ένταξη είναι 25 εκατομμύρια. Πολλά κράτη ζήτησαν έκτακτη βοήθεια. Η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος μεταξύ άλλων για 23,1 συνολικά. Έχουμε και άλλες βεβαιτήσεις που εξετάζουμε και αξιολογούμε βάσει των κριτηρίων που έχουν ήδη καθοριστεί. Η εμπειρία του 2014 είναι μια καλή εμπειρία. Όπου να ξεκινάμε με την επόμενη χρονιά. ελπίζω, μάλλον είμαι σίγουρη, ότι θα σας ενημερώσουμε και για τα προγράμματα εργασίας για το 2015 χωρίς άλλο. Αυτά που σας είπα αφορούν το 2014. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ή σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σίγκαν. Πρώτα η κυρία Σίπελ έχει ζητήσει το λόγο από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω συγκεκριμένα και άμεσα να υποβάλω ερώτηση για το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό, αλλά για τον ορισμό του που σχετίζεται και με την ε, εφαρμογή του. Γιορτάσαμε χθε ε, τα 25 χρόνια από την πτώση του τύπου του Βερολίνου στη Γερμανία. Μέχρι τότε σκοτώνονταν πολύ ε, στα σύνορά μας ζητούσαν βοήθεια για να εγκαταλείψουν την Ανατολική Γερμανία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και για τα προγράμματα εσωτερικής ασφάλειας και για το πρόγραμμα άσυλο μετανάστευση που αναφέρεται διαρκώς όπου λέει ότι πρέπει να καταπολεμούμε τους ε, περατές και τους λαθρεμπόρους, τους εμπόρους ανθρώπων. Υπάρχει κάποιος ε, διαχωρισμός αφενός μεν ε, από για διακινητές, λαθροδιακινητές και ανθρώπους, εμπόρους ανθρώπων από την άλλη, δουλεμπόρους. Δεν είναι πάντοτε εγκληματικές οργανώσεις ή μήπως θεωρούμε ότι οι διακινητές δεν είναι εγκληματική ερώτηση. Και τρίτον, ένας ε, σύρος ο οποίος προσπαθεί να βρεθεί σε ασφαλή χώρα και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός διακινητή μπορεί να, να λάβει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θεωρείται ήδη εγκληματίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω την ε, παρέμβασή μου στις μεταναστευτικές πολιτικές εν για να το πω σύντομα. Στη φάση συζήτησης για την προετοιμασία του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, το Ευρωκοινοβούλιο επέμεινε πολύ για μια ισορροπία, θα έλεγα, ανάμεσα στο σεβασμό των πολιτικών ε, ε, ένταξης, θα έλεγα, και των πολιτικών ε, ασφάλειας ή ασφάλιση των συνόρων. Άκουσα πολλά πράγματα για την ασφάλεια στη δική σας παρέμβαση, ενώ πολύ λιγότερα όσον αφορά την ε, ενσωμάτωση ή την επανεγκατάσταση. Επίσης, σημαντικό είναι το θέμα της χρηματοδότησης δράσεων ε, στις τρίτες χώρες. Και εδώ έχω κάποιες αμφιβολίες όταν ακούω τις χώρες με τις οποίες από ό,τι φαίνεται γίνονται, συνάπτονται συμφωνίες, Αιθιοπία και Σουδάν. Εκστρατεία ενημέρωσης για τους κινδύνους ε, παράνομης μετανάστευσης στις χώρες αυτές, όταν ξέρουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες, τους λόγους δηλαδή για τους οποίους φεύγει ο κόσμος από εκεί, ε, νομίζω πως η ενημέρωση για τους κινδύνους λαθρομετανάστευση δεν έχει και πολύ νόημα γιατί στην ουσία η αναλλακτική του είναι ο θάνατος. Το ίδιο όταν δίνεται και παράδειγμα της Αλβανίας, της Ουκρανίας, του Μαρόκου όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων. Μα θέση, σε ποια πολιτική εντάσσεται αυτή η Γενική Διεύθυνση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ποια είναι η πραγματική συνέχεια που δίνεται στις δράσεις μας με βάση αυτήν την ε, ε, συνιστόσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, κάνατε λόγο για ενίσχυση των ε, δυνατοτήτων των κρατών μελών να εντοπίζουν καλύτερα τα μικρά σκάφη. Για ποιο λόγο γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος που πνίγεται στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή είναι κόσμος που δυνητικά είναι ε, ετούντες άσυλο. Δεν το λέω εγώ, το λέει η πατιαρμοστία για τους πρόσφυγες, ότι το 80 με 85% είναι ετούντες άσυλο. Και τελειώνω, Πρόεδρε, μην ανησυχείτε. 80 με 85% είναι δυνητικοί ετούντες άσυλο. Οπότε, τι κάνουμε για να σεβαστούμε στο πλαίσιο των συζητήσεων που κάνατε την πρόσβαση στο άσυλο. Και ποια επιμονή ποια μπορεί να δείξει η Κομισιόν ώστε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα στο άσυλο και οι δυνατότητες αίτησης ασύλου να γίνουν σεβαστές. Έπειτα, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Εξωτερικά Σύνορα. Ε, εδώ δεν ολοκληρώθηκε το αίτημά μας επί τη βάση των πληροφοριών που μας είχατε δώσει. Στόχο είχε αυτό το πρόγραμμα να γίνονται τεκμηριωμένες μελέτες και σταθερές πληροφορίες όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στην Κομισιόν για να παίρνει αξιόπιστες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη στο θέμα. Μας είχατε πει ότι αυτό το πρόγραμμα θα εντασσόταν στο πρόγραμμα του 2015 και θέλω να ξέρω τι έχει γίνει. Σας ευχαριστώ. Και τελευταίος ο μιλητής... Eh, η κυρία Τσέβαλος, τους πράσινους. Και για μένα είναι κάπως νέα όλα αυτά. Ε, όταν ε, βλέπω τα έγγραφα και ακούω τα όσα είπατε, προκύπτουν κάποια ερωτήματα. τι γίνεται όσον αφορά την αρρωγή σε περιπτώσεις καταστροφών. Μιλάτε για βοήθεια που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες κρίσεις όπου οι πρόσφυγες μπορεί να χρειάζεται να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα. Αλλά εάν κατάλαβα καλά, εδώ μιλάμε για χρήματα τα οποία πάνε σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Τώρα, όταν μιλάμε για ανακούφιση μετά από καταστροφές, ε, φαντάζομαι ότι πρόκειται για αρρωγή που δίνουμε σε άλλες χώρες εκτός Ένωσης. Δηλαδή, αν υπάρξει ε, πραγματικά ανάγκη. Μα δεν λέμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε για το, πρόληψη αυτών των καταστροφών. Τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να αποφύγουμε τις ε, καταστάσεις αυτές όπου ο κόσμος βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο προκειμένου να μεταναστεύσει. Οι πλημμύρες και οι καταιγίδες αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο και ε, μαζί και οι πρόσφυγες γιατί οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται αδύνατες. Επίσης βλέπουμε ένα σωρό συγκρούσεις που κάνουν τον κόσμο να φεύγει γίνεται προληπτική δουλειά επί τόπου, ώστε να αποφεύγονται αυτού του είδους οι καταστροφές που ως κατάληξη έχουν να δημιουργούν δύσκολη κατάσταση και στα σύνορα της Ένωσης και εντός των ευρωπαϊκών χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόρα Φεράρα από το EFTD ζήτησε επίσης το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ. Εγώ αναρωτιόμουν το εξής. Αν γίνονται έλεγχοι για την χρήση αυτών των κονδυλίων. Για να δούμε δηλαδή αν οι στόχοι οι οποίοι αρχικά έχουν τεθεί συμπίπτουν με τα, με, με τα αποτελέσματα. Εγώ είμαι Ιταλίδα και στην Ιταλία φτάνουν διάφορα χρήματα για τη μετανάστευση, το άσυλο, τους επαναπατρισμούς κτλ. Αλλά εξακολουθούμε να είμαστε σε επίγουσα κατάσταση και σε βαθιά κρίση. Γι' αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η στόχη είναι κατάλληλη. Ε, μάλλον στα λόγια είναι κατάλληλη στόχη, αλλά πρέπει να δούμε αν γίνεται επαλήθευση ανάμεσα στους στόχους που αρχικά είχαν τεθεί και τα αποτελέσματα που τελικά επιτυγχάνονται ή όχι. Σας ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος και το λόγο έχετε πάλι και εσείς κυρία Σιγκάν για να απαντήσετε και να κλείσετε με τα σχολιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που θα ήθελα μάλιστα να επαναλάβω από τα όσα είπα στην αρχική μου εισήγηση είναι ότι εδώ μιλάμε για ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2014 το οποίο όμως δεν μπορεί να το δούμε απομονωμένα, θα πρέπει να το δούμε συμπληρωματικά με τα κεντρικά, κεντρική ροή χρημάτων που πηγαίνει για τα εθνικά προγράμματα που τα ίδια τα κρατή-μέλη μας υποβάλλουν, έχουν ε, υιοθετηθεί από την Κομισιόν και θα εφαρμοστούν. Ε, και αυτά είναι τα εθνικά προγράμματα, ε, τα επταετή. Τα χρήματα αυτά λοιπόν δίνονται στα κρατημέλη, τα διαχειρίζονται τα κρατημέλη. Εμείς ε, αυτό που έχουμε στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας μας είναι ένα κομμάτι των χρημάτων το οποίο άμεσα διαχειριζόμαστε εμείς και που μας επιτρέπει να συμπληρώσουμε σε ορισμένα προγράμματα τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη μέσω των εθνικών τους προγραμμάτων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε το σύνολο τις προσπάθειες και να μπορέσουμε να εμπιστευτούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς θα εξασφαλίσουμε και θα παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία καθώς και θα την ελέγξουμε εκ των υστέρων έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία και στην εφαρμογή των πολιτικών μας. Να μην υπάρχει η δυνατότητα, ε, πιθανότητα μάλλον, όπου κάπου εστιάζουμε περισσότερο ή λιγότερο. Μάλιστα, Πολύ ισχυρό στόχο είναι η χρήση του νέου μηχανισμού πολιτική, διαλόγων πολιτικής, γιατί έχουμε ε, διαλόγους για όλα τα μέσα και τα κονδύλια. Είχαμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη και να τους δείξουμε πως ε, διάφορες προτεραιότητες για τις πολιτικές μας ε, πρέπει να βρουν το χώρο τους στα εθνικά προγράμματα. Εάν δεν υπάρχει εκεί χώρος θα γίνει μέσα στο πλαίσιο των, εθνι... των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας αλλά πρέπει να επικρατεί μια γενική ισορροπία ώστε να ανταποκριθούμε στις ε, σημαντικές προτεραιότητες. Σας έδωσα κάποια παραδείγματα για, για τα προγράμματα και τις δράσεις του 2014 και λόγω αυτών των παραδειγμάτων, ε, ε, μάλλον εκτός από αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν και άλλα στα κείμενα, να σας στείλω το κείμενο, μπορώ να σας το στείλω. Είναι διαθέσιμα βέβαια και στο ίντερνετ. Μπορείτε να δείτε ακριβώς για ποιες δράσεις πρόκειται, καθώς και για τα ακριβή ποσά και μετά να το συζητήσουμε. Ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα μόνο, δεν ήθελα να σας δώσω την εντύπωση ότι μόνο αυτά κάνουμε. Ακολουθούμε τον ορισμό για την εμπορία ανθρώπων και για το λαθρεμπόριο δεν τα συγχαίουμε όλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία είναι μόνο στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Τα συζητάμε όπως και για άλλα θέματα, όπως σε όλες οι σημαντικές πτυχές για την ένταξη των, των, των άσυλων στα εθνικά προγράμματα. Πρέπει δηλαδή να τα δούμε αυτά όλα πολύ ρεαλιστικά. Για τα μέσα επίγουσες ε, ανάγκης, έκτακτης ανάγκης, αυτά έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρινόμεθα σε επίγουσες καταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν ήδη ε, και είναι κάτι τα διαφορετικά από την μόνιμη διαδικασία που έχει στόχο να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αυτό γίνεται μέσω της εφαρμογής των προτεραιοτήτων στα εθνικά προγράμματα. Οι μηχανισμοί της ανάγκης είναι πολύ σημαντικοί για έκτακτες περιστάσεις, αλλά δεν μπορούν να αντακαταστήσουν έναν μακροχρόνιο προγραμματισμό και μια μακροχρόνια διαδικασία που θα πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη οι ενημερωτικές εξαρτήσεις που κάνουμε στο πιλωτικό πρόγραμμα το ανέφερα γιατί είναι μία από τις πρώτες περιπτώσεις που κάνουμε κάτι τέτοιο. Αν δείτε την πολιτική για την παγκόσμια μετανάστευση και κινητικότητα. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες, χώρες προέλευσης ή διέλευσης. Μέχρι στιγμή δεν κάναμε κάτι τέτοιο, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα από τα πρώτα μας προγράμματα, θα το αξιολογήσουμε, θα το εκτιμήσουμε όπως και όλες οι άλλες δράσεις ε, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας και θα εξετάσουμε αν έφερε αποτελέσματα ή όχι. όσο για το το, το, την πτώση του τείχου του Βερολίνου ήταν πολύ ωραίο ο εορτασμό τη Εποτίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό όταν μιλάμε για ολοκλήρωση. Σα ευχαριστώ και εγώ σα ευχαριστώ που μα θυμήσατε του εορτασμού. Να επαναλάβω τα λόγια του Μάρτιν Σούλτ, του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου μα, ότι πρέπει να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε πολύ καλά και να φροντίσουμε ώστε να μην χτιστούν νέα τείχη γύρω από την Ευρώπη και μετά να πρέπει ξανά να το ε, Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τα όσα μας είπατε, για τα ενημερωτικά που μας είπατε για τα προγράμματά σας. Να τονίσω επίσης πως ε, πρόκειται για τα κοινοτικά προγράμματα και για τα κονδύλια για την μετανάστευση, την ολοκλήρωση και την ασφάλεια. Ε, το Δεκέμβριο θα ακούσουμε και για τα εθνικά προγράμματα και την κατάσταση πρόοδο, οπότε θα παρακολουθήσουμε, ε, θα έχουμε μάλλον συνέχεια όλων αυτών και σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. colleagues, um, the next point on the... Ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση των κύριων χρηματοδοτήσεων δύο μελετών υπό τον χώρο της Συνθήκης Λισαβόνας για το Γραφείο του Ευρωπαίου Σαγγελέα εξυγχρονισμό Eurojust Europol, σχέδια κανονισμών σχετικά έχουμε ενώπιον της Επιτροπής. Στόχος μας είναι ο κανονισμός να καλύψει και να, να διορθώσει κατευθύνσεις για τη συνεργασία στον χώρο της ποινικής δικαιοσύνης και της επίβολης του νόμου. Και έτσι ζητήσαμε αυτές οι δύο μελέτες για την υφισταμένη και μελλοντική συνεργασία μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών να μας παρουσιαστεί από τους δύο πυρογνώμονες που έχουν συντάξει τις σχετικές έρευνες. Έχουν διανεμηθεί τα κύρια σημεία των εκθέσεων. Καλώς ορίζω τις δύο στάκτρες. Ευχαριστώντας τες. Um, to my left uh, η κυρία Άννα Βάινμπεργκ, καθηγήτρια Άννα Βάινμπεργκ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκών Σπουδών στην, ε, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Και ο καθηγητής Πολ Ντεχερτς. Διευθυντής της Ομάδας Ερευνών Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Συνταγματικών κρατικών δομών, διευθυντής του τμήματος διατομεακών μελετών του δικαίου τον, του Φράι Universität Brüssel και δίνω τον λόγο παρακαλώ πρώτα εσείς κυρία Βάινμπεργκ Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μας αναθέσατε αυτή τη μελέτη για τη σχέση μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Η Νεφερμαντά και η Κλωέ με ε, στήριξαν στην ε, διατύπωση, στην κατάρτιση αυτών των εκθέσεων. Θα ήθελα ιδιαίτερως να ευχαριστήσω όλους τους ειδικού και τους ε, εκπροσώπους του κλάδου από τους οποίους πήραμε συνέντευξη. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές αποκεντρωμένες υπηρεσίες και φορείς στο χώρο, στον νέο χώρο δικαιοσύνης και ασφάλειας ε, που εμπίπτουν στις, ε, στον τομέα αυτής της ε, έρευνας, η οποία εστιάστηκε στη σχέση μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών για τις εξής υπηρεσίες, τη Europol, τη Eurojust, Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Απάτης και το ε, μελλοντικό γραφείο ε, δημοσίου κατηγόρου. Συνεργασία λοιπόν και διάρθρωση, σωστή διάρθρωση των εργασιών ε, μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών θα είχε πολύ μεγάλη σημασία για μια πολυτομεακή προσέγγιση για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την εγκαθιδρυσία ενός ασφαλούς χώρου δικαιοσύνης. Ωστόσο, επικάλυψη εργασιών και σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τομέων δραστηριοποίηση των υπηρεσιών μπορεί να υπάρχουν, χωρί αυτό να σημαίνει ότι πάντοτε είναι μειονέκτημα, μπορεί ακόμα και πλεονέκτημα να συνιστούν. Όταν όμω υπάρχει επικάλυψη, είναι απαραίτητη η ομαλή συνεργασία. Απαιτεί οι εμπλεκόμενε υπηρεσίε και φορεί να συνεργάζονται ε, χέρι με χέρι για να σέβονται, και να σέβονται το είναι εντολή η μία τη άλλη και, και να αξιοποιούν τι εμπειρίε του. Μια σειρά από εμπόδια όμως ε, έχουμε εντοπίσει. Καταχάζεται ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και φορέων, επειδή προέρχονται από διαφορετικές ε, γενναίες, άλλες έχουν μεγάλη πείρα, άλλες ακόμη αγωνίζονται να δικαιολογήσουν την προσθεμένη αξία που προσφέρουν. Ε, αγωνίζονται για διαφορετικούς στόχους η λογική καλύτερα, μια υπερεθνική λογική, η OLAF και η PPO, το γραφείο δηλαδή του Ευρωπαίου κατηγόρου, ενώ διακυβερνητική περισσότερο για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, τη Eurojust και τη Europol, που προσφέρουν υπηρεσίες. Έχουμε επίσης διαφορετικές ε, παραδόσεις από τους ε, που εκπροσωπούνται μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες. Eurojust, EGN, Europol είναι δικαστικά όργανα, η Europol είναι αστυνομικό όργανο και ούτω καθεξής. Διαφορές υπάρχουν ως προς τις δομές τους επίσης, αλλά και ως προς τους πόρους και τον προπολογισμό τους. Επίσης, διαφορές μεταξύ των εθνικών ποινικών συστημάτων ή συστημάτων δίωξης του εγκλήματος ε, εμπεριέχονται και εκφράζονται μέσα από την λειτουργία αυτών των υπηρεσιών το γεγονός ότι η, τα καθήκοντα και η λειτουργία του εις Βρετανικής Αστυνομίας στον Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαφορετικά από αυτά της Γαλλικής Αστυνομίας έχει, συνεργα... έχει συνέπειες ως προς τη συνεργασία της Europol και της Eurojust. Ε, βλέπουμε λοιπόν να απουσιάζει μια ενιαία θεώρηση της ε, ευρωπαϊκής ποινικής δικαιοσύνης γιατί και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει και υπηρεσίε χειρίζονται τα σχετικά θέματα, τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο. Προσωπικέ επαφέ και σχέσει μεταξύ μελών του προσωπικού των διαφόρων ευρωπαϊκών υπηρεσιών και σωμάτων, φορέων γενικότερα, και οι σχέσει αυτών με τι αντίστοιχε γενικέ διευθύνσει και τα εθνικά σώματα είναι πολύ σημαντικέ, ώστε να επηρεάζεται προ το ωφέλιμο η δουλειά αυτών των υπηρεσιών το νομοθετικό πλαίσιο εν τέλει έχει πολύ περιορισμένες διατάξεις και περιθώρια συνεργασίας, προβλέπει περιθώρια συνεργασίας πολύ περιορισμένο. Έτσι λοιπόν στην πρακτική η συνεργασία με τον μεταξύ των υπηρεσιών αυτών αναπόκειται στις ίδιες τις υπηρεσίες. Ο στόχος της μελέτης μας είναι να αναλύσουμε την κατάσταση και πιθανές εξελίξεις στη σχέση μεταξύ των υπηρεσιών για να εντοπίσουμε βέλτιστες πρακτικές, δυσκολίες και ενδεχομένω να προτείνουμε ε, στόχους βελτίωσης. Η μελέτη, η μελέτη χωρίζεται σε δύο τμήματα. Η μία αφορά τη συνεργασία μεταξύ των ε, υπηρεσιών για την ε, καταπολέμηση σοβαρού δεσυνοριακού εγκλήματος και η άλλη αφορά την, τον τομέα των λεγόμενο PIF. Έχουμε λοιπόν τις ε, σχέσεις της Europol με την ε, EGN και αντίστοιχα της ε, Eurojust με την Europol. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτές και τη δημιουργία του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κατηγόρου. Καταρχάς για την Europol και την Eurojust. Η Europol και η Eurojust έχουν και πολλά κοινά σημεία, αλλά και πολλέ διαφορέ. Ε, η Europol θεσπίστηκε με τον τρίτο πυλώνα του Μάστριχτ, έχει ιεραρχική δομή και καθοδήγεται από τις αρχές της επιβολής του νόμου και τον πρακτικό ρεαλισμό, ενώ η Eurojust θεσπίστηκε αργότερα από τον τρίτο πλήνο του Άμστερνταμ, έχει συλλογική δομή και πολύ ε, έντονο δικαστικό χαρακτήρα, με διαφορετικούς βέβαια πόρους Παρά το γεγονός αυτό, είναι η Europol και η Eurojust αδελφές υπηρεσίες. Έχουν κοινό πεδίο ουσιαστικά αρμοδιοτήτων, δηλαδή την καταπολέμηση του διεθνικού ή διασυνοριακού εγκλήματος και έχουν παρόμοια σχέση κάθε μία τους με τις εθνικές αρχές. Οι εθνικές αρχές παραμένουν δηλαδή οι κύριοι και οι κάτοχοι της ποινική δίωξης ανάκριση και δίωξη. Και έτσι μόνο οι υπηρεσίε μπορούν να προσφέρουν η Europol και η Eurojust στι εθνικέ αρχέ. Σε εθνικό επίπεδο. Η συνεργασία μεταξύ των ε, αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν πολλοί συγκριτισμοί μεταξύ των δύο υπηρεσιών με νομικούς όρους. Λίγες ε, διατάξεις προβλέπουν ε, συγκεκριμένα νομοθετικά μέσα για την Europol και την Eurojust. Υπάρχουν κάποιες περιστορές ε, ιδέες μέσα στις προτάσεις και τις διαπραγματεύσεις. Η δεύτερη δε συμφωνία συνεργασίας που θα σπίσει το 2010 μεταξύ Europol και Eurojust αποτελεί το κύριο μέσον, κύριο εργαλείο που διέπει τις σχέσεις τους. Στην πράξη, η διμερή συνεργασία έχει αναπτυχθεί και βελτιωθεί σε σύντο χρόνο. Στενή και τακτική συνεργασία περιγράφουν αρκετές κοινέ πρωτοβουλίε και επιτυχής, επιτυχή εγχειρήματα και η δυνατότητα ιδιαίτερως στην συνεργασία για την επιτύχηση κοινών στόχων. Αλλά παραμένουν κάποια προβλήματα. Ιδιαίτερα έχουμε εντοπίσει τέσσερα κύριε το πρώτο αφορά το συντονισμό των δικαστικών αρχών. Με βάση τη συνθήκη, η Eurojust συντονίζει τις δικαστικές αρχές, ενώ η Europol συντονίζει τις αρχές επιβολής του νόμου. Ωστόσο, στην πράξη, η κατανομή των καθηγόντων... αλλά στην πράξη, ιδιαίτερα μέσα στη διαδικασία των ανακρίσεων, είναι πολύ περίπλοκη αυτή η κατανομή των αρμοδιότητων και λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα των ε, εθνικών ποινικών συστημάτων. Άρα χρειάζεται μια κάποια ευελιξία και από αυτήν προκύπτουν γκρίζε ζώνε. Όπου μπορεί η, ο διαχωρισμό των αρμοδιότητων μεταξύ των δύο υπηρεσιών ασφαλώ να, να, να, να εμφανίζεται δύσκολο και αυτό οδηγεί σε εντάσει μεταξύ των υπηρεσιών. Εντάσει οι οποίε είναι ιδιαίτερως αισθητέ λόγω της ε, διατύπωσης μιας διάταξης στη Γενική Προσέγγιση του Συμβουλίου στον κανονισμό για τη Europol, όπου ορίζεται ότι θα συντρέχει τις εθνικές αρχές ε, επιβολής του νόμου, τις ευρωπαϊκές, η Europol, αλλά και άλλες αρχές εν γέννη. Εν προκειμένου δεν υποστηρίζουμε μια αυστηρή, έναν αυστηρό διαχωρισμό ε, τυπικό διαχωρισμό αρμοδιότητα μεταξύ Europol και Eurojust, διότι αυτό θα επιβάρει ιδιαίτερα την ευχέρεια και την ευελιξία που θα μπορούσαν να έχουν στη θέση τους οι εθνικές αρχές. Αλλά επιμένουμε ότι θα πρέπει η κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπεται από τι συνθήκες να γίνεται σεβαστή. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το γράμμα του άρθρου 88 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια διάταξη επίσης θα πρέπει να προσθεθεί και στους δύο κανονισμούς. Μια διάταξη η οποία θα υπογραμμίζει την υποχρέωση της κάθε μίας από τις υπηρεσίες αυτές ε, να σέβεται την ε, ύπαρξη και την ε, λειτουργία και το κύρος της άλλης. Δεν θα έχω βέβαια το χρόνο να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες που θα ήθελα. Θα επανέλθω όμως αργότερα αν το θέλετε. Το δεύτερο θέμα αφορά τις ε, κοινέ ομάδες ε, ερευνών. Ξέρετε ότι πρόκειται για μεικτό μέσον, στο οποίο έχουμε και επιβολή του νόμου και δικαστικές αρχές. Έτσι λοιπόν, λογικό είναι η Europol και η Eurojust να υποστηρίζουν τις κοινέ αυτές ομάδες, αλλά με διαφορετικό ρόλο. Αυτέ οι τζίτι, κοινέ ομάδε ερευνών, Πολλέ φορέ πολύ συχνά αναφέρονται σαν καλό παράδειγμα συνεργασία μεταξύ Europol και Eurojust. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν εντάσει. Και κυρίω λόγω τη δυσκολία στη χρηματοδότηση και από τα δύο σχέδια κανονισμού. Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα από την επικάλυψη. Γιατί θα προκύψει και περισσότερο, περισσότερο δυνατότητα για χρηματοδότηση για τις κοινέ ομάδες ερευνών. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος οι εθνικέ δικαστικές αρχές να περιθωριοποιηθούν γιατί οι κοινέ αυτές ομάδες θα έχουν προσθέτει δυνατότητα χρηματοδότηση και θα έχουν και διπλή ακόμα χρηματοδότηση Europol και Eurojust. Πιστεύουμε ότι, ένας ότι θα χρειαστεί ένας μηχανισμός για την αποφυγή διπλή χρηματοδότηση και ίσως μια υποχρέωση αμοιβαίας ενημέρωση να αρκεί για να αποφευχθεί αυτό. Όπως επίσης και η θέσπιση μιας κεντροποιημένη υπηρεσία που θα διοχετεύει τα σχετικά αιτήματα. Επιπλέον υπάρχει ανάγκη να διευθετηθεί η ανισότητα στις διαθέσιμες Europol και Eurojust ε, δυνατότητες χρηματοδότησης. Επίσης, τρίτος τομέας, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Europol και Eurojust, που έχει περιπλακεί ή έχει υπάρξει περίπλοκη στο παρελθόν λόγω της ε, αρχής του κατόχου owner principle, βάση της οποίας μόνο ο κύριος που κατέχει την πληροφορία αποφασίζει αν θέλει και πώς να την διαβιβάσει. Στο παρελθόν τα κράτη απέφευγαν να διαβιβάσουν από τη Europol στη Eurojust πληροφορίες. Τώρα βλέπουμε ότι σημειώνεται βελτίωση. Επί παραδείγματι η Eurojust σχετίζεται, συνεργάζεται με πολλά από τα ε, κέντρα της Eurojust. Αλλά χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη της αλλαγής πληροφοριών και εισάγονται δύο συναφείς διατάξεις που συνεπάγονται ε, το λεγόμενο αντικατοπτρισμό, δηλαδή την αντανάκλαση μιας πληροφορίας στα συστήματα πληροφοριών, από το ένα σύστημα πληροφοριών στο άλλο. Τέτοιο και τελευταίο θέμα που εντοπίζουμε, η ανάλυση της πληροφορίας για λειτουργικούς και στρατηγικούς στόχους που πάντα βρισκόταν στο επίκεντρο της εντολής της Europol πρόσφατες εξελίξεις τις αναλυτικές, το αναλυτικό δυναμικό της Eurojust, λειτουργικό και στρατηγικό, οδηγούν σε ανησυχίες ότι μπορεί να υπάρξει επικάλυψη έργου λόγω ομοιότητας των δραστηριοτήτων. Αλλά μια πιο προσεκτική ανάλυση μας λέει ότι η Eurojust έχει ανάλυση περισσότερο δικαστικού προσανατολισμού και της Europol η ανάλυση έχει διαφορετικό προσανατολισμό και άρα χρειάζεται η λεγόμενη διαπαιδαγώγηση, λεγόμενη παιδαγωγική προσπάθεια, ώστε να υπογραμμιστούν οι σαφείς διαφορές που υπάρχουν. Και τώρα θα περάσω στο δεύτερο τμήμα της πρότασής μας για να, και θα περάσω κατευθείαν στην ε, δημιουργία της υπηρεσίας του Ευρωπαίου Κατηγόρου. Η θέσπιση ενός Ευρωπαίου Κατηγόρου θα επηρεάσει ασφαλώς τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και φορέων που εργάζονται στον χώρο αυτόν. Αλλά πρόωρα στάδια των διαπραγματεύσεων εμποδίζουν λεπτομερή ανάλυση πιθανή συνεργασία μεταξύ του Γραφείου του Ευρωπαίου Κατηγόρου και των ε, ομολόγων. Βέβαια, όσον αφορά τον ορισμό της ειρήνης και για το πόσο το ΙΠΠΟ έχει αποκλειστικές ή κοινέ αρμοδιότητες. Δεύτερον, το η δομή του ΙΠΠΟ που θα, και ξέρετε ότι πάμε προς μια συλλογική δομή του ΙΠΠΟ και τρίτον, ο αριθμός των ε, συμμετεχόντων μελών. Τώρα όσον αφορά τις πιθανές σχέσεις ανάμεσα στο ΙΠΠΟ στον Ευρωπαίο κατήγορο και το Eurojust, ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ενώ και τα δύο σώματα έχουν κοινή δικαστική λογική, αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης. Το πιο λεπτό θέμα είναι ίσως η ακριβής έννοια της ε, έκφρασης από την Eurojust που όπως αυτή ονομάζεται ε, αναφέρεται στο άρθρο 16 της συνθήκης. Σύμφωνα με την πρόταση της ε, Κομισιόν, ο Ευρωπαίος Συνήγορος βασίζεται στο γεροντάζ για διοικητικά και διαχειριστικά θέματα και αυτό υποτίθεται ότι θα γίνει με μηδενικό κόστος. Ε, η Eurojust όμω έχει εκφράσει την ανησυχία της για το πώ θα το πετύχει αυτό, χωρί να θέτει σε κίνδυνο τι δικέ τη δραστηριότητε. Η τοποθεσία, η έδρα του Ευρωπαίου κατηγόρου ε, είναι άγνωστη και ε, η πρόταση αυτή θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να υλοποιηθεί αν ο Ευρωπαίος κατήγορος δεν εγκατασταθεί στην Χάγη. Έχουμε τρία δυνατικά μοντέλα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά φυσικά μπορούμε να τα ε, συζητήσουμε αργότερα. Υπάρχει επίσης μια δυνατότητα ε, δημιουργίας μιας πιο διαφορετικής σχέσης ανάμεσα στον κατήγορο και στο Eurojust. Για παράδειγμα, τα εθνικά μέλη του Eurojust θα μπορούσαν να γίνουν Ευρωπαίοι εισαγγελείς ή αντισεγγελής, Αλλά αυτό θα είναι πιο δύσκολο. Ή ο δημόσιος κατήγορος θα μπορούσε να συνδέεται με το συλλογικό όργανο της Eurojust. Επίσης, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει ανάγκη να σκεφτούμε την επιχειρησιακή συνεργασία στην πράξη, γιατί το Eurojust ούτως ή άλλως θα εξακολουθήσει να παίζει ρόλο ε, μετά από την ε, ε, εγκαθίδρυση του Ευρωπαίου κατηγόρου. Τώρα, όσον αφορά τον κατήγορο και την Όλαφ. Και αυτό το θέμα ε, προκαλεί διάφορα ζητήματα, όπως το μέλλον της Όλαφ. Η Όλαφ ε, μάλλον θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Όμως, το τμήμα του προσωπικού της θα μπορούσε να μετακινηθεί υπό τον κατήγορο. Η συνεργασία ανάμεσα στους δύο σίγουρα θα συγχρειαστεί. Για παράδειγμα, στον τομέα της ανάλυσης πληροφοριών. Για την ώρα όμως η μόνη διάταξη προς αυτό το σκοπό στην πρόταση της Κομισιόν για τον κατηγόρο είναι αρκετά αόριστη και βασικά αναφέρεται στο συμπέρασμα μιας, στην μάλλον στη σύναψη μιας συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στους δύο. Τώρα, κατήγορος και Europol. Και εδώ θα χρειαστεί βεβαίως σε συνεργασία. Ωστόσο και πάλι η πρόταση της Κομισιόν είναι αρκετά όριστη και μόνο αναφέρεται σε μια ειδική σχέση ανάμεσα στους δύο που συμπεριλαμβάνει και την ανταλλαγή πληροφοριών. Δυστυχώς είναι πολύ νωρίς για να μπούμε σε λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα, γιατί όλα αυτά θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές που θα πρέπει να γίνουν σε σχέση με τον ε, δημόσιο κατήγορο. Πριν να κλείσω λοιπόν, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη να εξεταστεί η πιθανότητα αναβολή τη διαπραγμάτευση και τη υιοθέτηση των διατάξεων που σχετίζονται με τη σχέση ανάμεσα στα υφιστάμενα ε, σε οργανισμούς και σώματα και τον ε, κατήγορο μέχρι ότου ο τελευταίο να πάρει την τελική του μορφή. Ε, ίσως εδώ και πάλι όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να αποφεληθεί της διαδικασίας ε, συναπόφασης ή αλλιώς αυτά τα θέματα θα πρέπει να ε, τα αποφασίζονται με ένα πιο οριζόντιο κείμενο όσον αφορά τις δύο, ε, οργανισμές, ε, διοργανικές σχέσεις στο τομέα του ΠΙΦ, στο πλαίσιο του ΠΙΦ, ώστε να υπάρχει εδώ συναπόφαση. Συμπεράσματα. Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών είναι εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, ειδικά στο, πλαίσιο, στο ισχύον πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η ευκαιρία αυτή θα πρέπει να γίνει λαμπή για να διευκρινιστούν διάφορα στοιχεία και να προχωρήσουμε σε μια πιο συνεχή, συνεπή ε, διαδικασία, έτσι ώστε να αποφευθούν τα εμπόδια αλλά και το αγωνισμό για τη συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα σώματα. Μπορούμε να επιμείνουμε όσον αφορά τη σημασία τη αμοιβή αμοιβαία γνώση, αμοιβαίων επαφών και κατάρτισης στην Ένωση και στο εθνικό επίπεδο, ώστε να μειωθεί η σύγχυση και οι εντάσει. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εδώ πολύ βασικός, γιατί είναι το καλύτερο βήμα ώστε να υπάρξει μια συνολική και συνεπής ε, εικόνα για τον ε, χώρο, τον ευρωπαϊκό χώρο ποινικής ποινικού δικαίου και επίσης θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να ισχύσει η απαραίτητη ε, ισορροπία ανάμεσα στην επιβολή του νόμου και τις δικαστικές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ασχοληθεί με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχέσεων ανάμεσα στους οργανισμούς, για παράδειγμα, ε, ε, καλώντας τους διάφορους επικεφαλείς των οργανισμών ε, στη Κοινοβούλιο την ίδια μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η πρώτη μελέτη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών στον τομέα της επιβολής του νόμου. Τώρα έρχομαι στην δεύτερη μελέτη για το καθεστώς προστασίας δεδομένων και την μελλοντική αρχιτεκτονική του τομέα της επιβολής του νόμου. Θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Ντεχέρτ. Δέκα λεπτά έχετε κι εσείς. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στα αγγλικά θα μιλήσω κι εγώ. Έχω ετοιμάσει κάποιες διαφάνειες εξάλλου στα αγγλικά. Ποιος είναι ο ρόλος μου εδώ σήμερα. Είναι να συζητήσουμε για την προστασία δεδομένων. Ό,τι πτυχές σχετικές με την προστασία δεδομένων έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη και την επιβολή του νόμου. Α, εδώ βλέπετε το όνομά μου. Λοιπόν, κατακαιρματισμός είναι κάτι βασικό και συνεχής μεταρρύθμιση σε όλα τα επίπεδα. Κατακαιρματισμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό του πλαισίου της προστασίας δεδομένων. Όπως είδαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση, ισχύει και εκεί αυτό, αλλά ισχύει και εδώ, ότι υπάρχουν διαφορετικά νομικά πλαίσια. Και δεν υπάρχει εναρμόνιση, ούτε καν συμβατότητα πολλές φορές. Επίσης υπάρχει μια συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο μου και των νομικών κειμένων όλων αυτών των οργανισμών για την προστασία των δεδομένων αλλά και σε υψηλότερο επίπεδο υπάρχει μεταρρύθμιση για τις προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν. Είτε πρόκειται για την οδηγία που θα γίνει κανονισμός, είτε πρόκειται για την απόφαση πλαίσιο όσον αφορά την προστασία δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου που θα γίνει οδηγία. Άρα λοιπόν υπάρχει μεταρρύθμιση σε δύο επίπεδα. Εγώ προσωπικά δεν προτείνω οι δύο αυτές λέξεις κλειδί που είναι ανησυχητικές. Μας συνόδευαν πάντα. Να ξέρετε ότι από μόνες τους δεν είναι το κακό. Το ερώτημα όμως σήμερα τίθεται. Όταν έχουμε αυτή την κατακαιρματισμένη εικόνα, αν τύχει καλής διαχείρισης, έχουμε μια καθαρή εικόνα για το τι πρέπει να κάνει κανείς όταν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Εγώ θα έλεγα όχι. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο κατακαιρματισμός είναι τόσο μεγάλος που επηρεάζει τη διαφάνεια και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ένα δεύτερο στοιχείο που μας οδηγεί στο να συμπεράνουμε ότι επιγόντως πρέπει κάτι να κάνουμε, αυτό είναι ότι το άρθρο 16 της Εθνικής Ήδης Ευρωπαϊκής Ένωσης επιμένει στην ανεξάρτητη μεταρρύθμιση όλων όσων έχουν να κάνουν με την προστασία των δεδομένων. Εμένα βέβαια εντάξει, πολύ μου αρέσουν όλα τα κείμενα για την προστασία δεδομένων στα κείμενα της Europol, της Eurojust και αλλού. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο λείπει. Και αυτό είναι η ανεξαρτησία και η εποπτεία. Πέρα δηλαδή από το επιχείρημα ότι είναι κατακαιρματισμένη η κατάσταση, υπάρχει και ένα άλλο πιο νομικό επιχείρημα που μας οδηγεί στην αναγκαιότητα κάτι να κάνουμε για να μπορούμε να σεβόμαστε το άρθρο 16 της συνθήκης. Τώρα, το κατεπήγον. Όταν δούμε αυτά τα κείμενα καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει πολλή δουλειά, υπάρχει πολλή πολιτική σοφία υπάρχει ανησυχία για την αποτελεσματικότητα της επιβολής του νόμου, όλα αυτά υπάρχουν. Αν όμως δούμε την ανταλλαγή πληροφοριών που γίνεται μεταξύ οργανισμών ή με τρίτα μέρη, με τρίτες χώρες, τότε οπωσδήποτε πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα τι ισχύει. Και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και για μένα ήταν μια σημαντική προσπάθεια γιατί μπορεί σε έναν οργανισμό να υπάρχουν καλές ρυθμίσεις που ρυθμίζουν την ε, μεταβίβαση δεδομένων κτλ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το καυτό ερώτημα που λέει ποιος εποπτεύει την ε, μεταβίβαση αυτή δεδομένων. Για μένα πρέπει να υπάρχει μια σαφής απάντηση στην ερώτηση. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ασχολείται με το νομικό πλαίσιο σήμερα πρέπει να το κάνει όχι μόνο στατικά, για το πώς δηλαδή ο κάθε οργανισμός επεξεργάζεται τα δεδομένα του, πιο δυναμικά, δηλαδή όταν ανταλλάσσονται αυτά τα δεδομένα, ποιος το υποπτεύει αυτό. Αυτή η πιο δυναμική προσέγγιση των ανταλλαγών μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών ή μεταξύ ευρωπαϊκών οργανισμών και τρίτων μερών και κυρίως με χώρες που δεν έχουν νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, αυτό είναι που μας προβληματίζει είτε πρόκειται για εντάλματα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Εκεί είναι που πρέπει να δούμε πού θέλουμε να πάμε όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Και ότι η επιβολή του νόμου ε, επιβάλλει και σε όσους ασχολούνται με αυτήν να τηρούν το απόρριτο για τα προσωπικά δεδομένα, ξέρουμε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται πάντα. Η προστασία δεδομένων, δηλαδή, είναι κάτι που χρειάζεται επιπλέον από το απόρριτο το οποίο είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όσοι υπηρετούν την επιβολή του νόμου. Στην δικιά μας μελέτη λοιπόν τι κάναμε εμείς. Συζητήσαμε αυτό το κατακαιρματισμένο πεδίο εκφράζοντας την ανησυχία μας και συζητήσαμε και την ανάγκη που υπάρχει για ανεξάρτητη εποπτεία. Υπάρχουν ε, όργανα που σε ένα βαθμό το κάνουν. Αυτό που μας απασχόλησε μας είναι η συμπληρωματικότητα των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία γιατί δεν είναι δυνατόν να απομονώσουμε το ένα όργανο από το άλλο. Αυτά λένε οι πρώτες σελίδες της μελέτης μας που έγραψα και που ελπίζω να διαβάσετε. Έπειτα περνάμε στα σενάρια. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτό το κατακαιρματισμό. Το πρώτο μου μήνυμα είναι όχι πανικός. Πολλά από τα σενάρια και τα πιο ρεαλιστικά εξελίσσονται έτσι ώστε να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εποφεληθεί από το χρόνο και να προχωρήσει βήμα-βήμα. Εντοπίσαμε λοιπόν διάφορα σενάρια και το πρώτο είναι να, να θεωρήσουμε το σχέδιο οδηγίας και να αποτελέσει στοιχείο αναφοράς που να περιλαμβάνει όλες τις προδιαγραφές για κάθε διαδικασία και δραστηριότητα που έχει να κάνει με την επιβολή του νόμου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ περιλαμβάνουμε και την επεξεργασία δεδομένων από, τις, από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Μπορεί να είναι βέβαια ιδεώδες σενάριο αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα νομικό σημείο αναφοράς μόνο. Και η διαφάνεια και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι κάτι που εξυπηρετείται έτσι πολύ καλά. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και υπάρχει και μια νομική ένσταση. Μπορεί κανείς με μια οδηγία να αντιμετωπίσει τις ρυθμίσεις στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τέτοιες λεπτομέρειες μερικές φορές έχουν τεράστια σημασία. Οπότε και αυτό το ιδεώδες σενάριο, αυτό σημαίνει ότι ό,τι κείμενα νομικά έχει αυτή τη στιγμή η Europol, η Eurojust για να ρυθμίζονται και άλλοι οργανισμοί, όλα αυτά θα μπουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο. Το δεύτερο σενάριο είναι το λεγόμενο segregated model, Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα. Κάποια πλεονεκτήματα υπάρχουν. Το κύριο είναι ότι είναι τόσες αλλαγές που πρέπει να γίνουν που αν δεν κάνουμε τίποτα, τότε στέλνουμε ένα μήνυμα προς αυτούς που ασχολούνται με τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων και τους λέμε ότι εσείς ασχολείστε με αυτό. Από την άλλη βέβαια δεν αντιμετωπίζεται έτσι το θέμα που λέει ότι πρέπει να έχουν περισσότερη δύναμη οι ίδιοι οι πολίτες όταν πρόκειται για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δεν προβλέπεται κάποια ανεξάρτητη αρχή εποπτείας. Το δεύτερο αυτό σενάριο, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα, αποδυναμώνεται από τα επιχειρήματα αυτά και δεν θα έπρεπε να το συμπεριλάβουμε σαν λύση. Υπάρχουν και άλλα δύο, το 3 και το 4. Αλλά δύο σενάρια, τα οποία είναι τα πιο πιθανά. Πολιτικά περισσότερο βιώσιμα. Το τρίτο σενάριο είναι εκείνο που λέει ότι θα ψηφίσουμε την οδηγία και θα βάλουμε ένα χρονικό όριο για την ε, αντικατάσταση και την προσαρμογή όλων εκείνων των κεφαλαίων στα διάφορα κείμενα που έχουν να κάνουν ε, με την προστασία δεδομένων στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Έτσι, κάποια στιγμή θα πάρει το πράσινο φως η οδηγία με ένα χρονικό ορίζοντα, οπότε υπάρχει χρόνος να γίνουν οι προσαρμογές που χρειάζεται. Ωραία. Πολύ λογικό αυτό. Θα πάρει χρόνο βέβαια για να συνηθίσουμε τη νέα αρχιτεκτονική προστασίας δεδομένων στη Γενική Οδηγία για την επιβολή του νόμου, αλλά και στο Γενικό Κανονισμό για όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων. Το θετικό είναι ότι μας προσφέρει χρόνο η λύση αυτή να προχωρήσουμε βήμα-βήμα και να συνηθίσουμε όλη αυτή τη νέα αρχιτεκτονική μέσω της οδηγίας και του κανονισμού που σας είπα. Ναι, λοιπόν. Καλό αυτό. Το αρνητικό ποιο είναι. Αν υποσχεθείτε, αν ψηφίσετε μια οδηγία και υποσχεθείτε να ξαναδείτε το όλο θέμα, τότε πάλι έχετε κολλήσει στην οδηγία. Και όπως είπα και πριν, η οδηγία δεν είναι το καταλληλότερο μέσο για να ρυθμίσει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Χρειάζεται κανονισμός. Εγώ δεν τα ξέρω όλα αυτά πάρα πολύ καλά, αλλά φαίνεται ότι έτσι ισχύει. η δικηγόρη, αυτό λένε. Χρειάζεται κανονισμός δηλαδή τελικά, δεν φτάνει η οδηγία. Και το άλλο είναι ότι αναθεωρώντας όλα αυτά τα κείμενα των ευρωπαϊκών οργανισμών, ό,τι ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων. Αυτή η τρίτη επιλογή που βάζει χρονικό ορίζοντα, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις, ότι τελικά θα περάσουν κάποια χρόνια. Μπορεί να μην είναι θεμελιώδες ζήτημα για σας, αλλά είναι κάπως περίεργο κάποιος να φτιάξει κάτι σήμερα ξέροντας ότι μετά από δύο χρόνια θα το αλλάξει. Τα δεδομένα. Πέρα αυτού δεν πρόκειται. Αυτό δεν είναι η Ευρώπη. Τέλος υπάρχει και ένα άλλο ενωπημένο, εναλλακτικό ενωπημένο μοντέλο, το τέταρτο σενάριο. προκειμένου να αναθεωρηθεί ο κανονισμός 45 2001, ο κανονισμός που έχουμε για τον Ευρωπαίο Επόπτη Δεδομένων, ο οποίος υποσχέθηκε αναθεώρηση του κανονισμού αυτού. Κάτι αναγκαίο, γιατί ο Ευρωπαίος Επόπτης Προσωπικών Δεδομένων στο μέλλον θα έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και στην διαδικασία υποβολής του νόμου. Έχει δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα ο Ευρωπαίος Επόπτης με τις νομοδοτήσεις του, με τις παρεμβάσεις του, αλλά ο κανονισμός 45 κάθετος 2001 δεν αναφέρει τίποτα για την επιβολή του νόμου. Πρόκειται για μέσο πρώτου πυλώνα. Άρα είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία αναθεώρησή του. Πολύ και στο Μοτεσκέ, γιατί τι είναι. Ψηφίζεται μια οδηγία αφήνετε όλους τους οργανισμούς με τις δικές τους νομοθεσίες και επανέρχεστε όταν αρχίζετε να προβληματίζεστε για ένα νέο κανονισμό 45-2001. Θα ήταν μια καλή εναλλακτική λύση. Υπάρχει πολύ σοφία μέσα σε μια τέτοια ρύθμιση, γιατί δίνει και χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι τότε θα έχετε δύο προδιαγραφές την οδηγία που θα ψηφίσετε τώρα και τον νέο κανονισμό για τον Ευρωπαίο επόπτη που θα ψηφίσετε στο μέλλον. Νομικά μιλώντας δηλαδή, μια τέτοια κατάσταση δεν είναι ιδεώδης. Ένα από τα δύο θα υπερέχει του άλλου, από αυτά τα δύο μέσα δηλαδή. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται και κάποια άλλα μικρά νομικά προβλήματα. Ένα θα ήταν ότι αν αναθεωρήσουμε το ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη Δεδομένων και έχουμε φτιάξει η ομάδα εργασία 29 κλπ. και αφήσουμε και τον ρόλο που έχουν οι εθνικοί επόπτες δεδομένων, πώς θα υπάρξει εναρμόνιση του ρόλου τους, των εθνικών δηλαδή εποπτών δεδομένων. Αυτό είναι μια δυσκολία που έχει το τέταρτο σενάριο, αλλά είναι κάτι που βρίσκουμε ενδιαφέρον. Έχω προσθέσει και δύο άλλες εναλλακτικέ που δεν είναι όμως τόσο πιθανές, την πέμπτη και την έκτη λύση. Να μην κάνουμε τίποτα με την οδηγία, να μην κάνουμε τίποτα με τον νέο κανονισμό για τον Ευρωπαίο Επόπτη. Ας μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Αυτό είναι λίγο, θυμίζει λίγο τη δεύτερη λύση που σας εξήγησα πριν, και η κριτική βέβαια είναι ακριβώς ίδια, ότι έτσι παραμένουμε σε μια κατακαιρματισμένη κατάσταση και δεν ανταποκρινόμαστε στο άρθρο 16 της συνθήκης που μιλάει για έναν ανεξάρτητο επόπτη. Και η τελευταία λύση είναι μια παραλλαγή του δεν κάνουμε τίποτα. Λέει ας προχωρήσουμε, ας αναθεωρήσουμε όλα τα κείμενα και ας αφήσουμε τον επόπτη βάσει του κανονισμού 45-2001 που ψηφίστηκε πριν από 10 χρόνια. Και ας αναλάβει αυτός το ρόλο του ανεξάρτητου επόπτη. Αλλά και εδώ υπάρχει η ίδια κριτική ότι δηλαδή δεν μπορείτε να πείτε ότι μια τέτοια ρύθμιση βάσει του κανονισμού 45-2001 καλύπτει τα όσα αναφέρει το άρθρο 16 της συνθήκης αφού δεν αναφέρεται η επιβολή του νόμου. Αυτά είχα να σας πω. Έξι σενάρια μελέτησα και το διασκέδασα. Πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα αυτό το κατακαιρματισμένο τοπίο στο όνομα των πολιτών. Ιδίω γιατί δεν πρόκειται μόνο για τη συλλογή δεδομένων αλλά και για την ανταλλαγή δεδομένων. Ποιος θα υποπτεύει όλα αυτά. Και ακριβώς εδώ είναι που έρχεται το άρθρο 16, το οποίο δεν έχουμε καλύψει μέχρι τώρα. Δεν, έχει, δεν μας έχει κοστίσει πολύ μέχρι τώρα, αλλά είναι ένα απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική εποπτεία και εσωτερικά και εξωτερικά. Προτείνω λοιπόν το κοινοβούλιο σας να εξετάσει καλύτερα τα έξι αυτά σενάρια. Επιμένω το άρθρο 16 μας επιτρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά με νέο μάτι. Μας επιτρέπει να έχουμε μια προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι ενιαίας αγοράς. Το άρθρο 16 δηλαδή μας επιτρέπει να ξεχάσουμε τους περιορισμούς της ενιαίας αγοράς. Η προστασία δεδομένων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κανένας αυτή τη στιγμή δεν έχει την συνολική εικόνα και εποπτεία και αυτό είναι το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Και τώρα μπορούμε να ακούσουμε τη συζήτηση. Να καλέσουμε τους συναδέλφους να δω, εδώ, να πούν τις σκέψεις τους, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στους εμπειρογνώμονες μας που είναι εδώ σε θέματα συνεργασίας. Δεν έχουμε κανένα έτοιμο προς το παρόν. Όσο να σκεφτείτε λοιπόν κάτι εσείς, θέλω να διατυπώσω μια ερώτηση προς το καθένα σας. Καταρχάς, για την κυρία Βάινμπερ και την πρώτη παρουσίαση. Αναφερθήκατε στο σημαντικό ερώτημα της θέσπισης από την Eurojust του, Ευρωπαϊκού, του, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κατηγορού και των συνοποιών αυτού. Και για μας είναι σημαντικό αυτό και να καταλαβαίνουμε επίσης και τι επιπλέον ευκαιρίες μπορεί να προσφέρονται στο πλαίσιο της Eurojust και της συνεργασίας. αλλά και πώς θα αλληλεπιδρούν η μία υπηρεσία με την άλλη. Αυτή την ερώτηση έχω για σας. Για τον ε, κύριο Τεχέτ μετά. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. είναι μια από τις πιο περίπλοκες διατυπώσεις που έχει και αυτή, η σχετική με το έργο της ε, Eurojust και την ερμηνεία, της, ερμηνεία του. Δεν βλέπετε τις εφάνειες. Γιατί στις διαφάνειες ε, παρουσιάζουμε τρία πιθανά μοντέλα να έχει το προπολογισμό, τη διαχείριση του προπολογισμού του δημοσίου κατηγόρου Eurojust. Και έτσι ο δημοσίος κατηγόρος να μην έχει χωριστό προσωπικό. Θα λέγαμε δύο κύκλοι ομόκεντροι. Με μεγαλύτερη τη Eurojust και μικρότερο κύκλο την ε, υπηρεσία του Ευρωπαίου Κατηγόρου. Διαφορετικά θα είχαμε δύο σώματα, δύο ε, χωριστές ε, δηλαδή οργανογράμματα και προπολογισμό. Αλλά όποτε έκανε δουλειά για τον δημόσιο κατήγορο η Eurojust θα αποζημιωνόταν. Άρα θα είχαμε διαφορετικούς κύκλους. Άλλα διάθεση των δυνατοτήτων της Eurojust στην IPPO. Και τρίτη λύση δύο χωριστά σώματα, προσωπικό και προπολογισμό, αλλά με κοινέ υπηρεσίε, επί παραδείγματι πληροφορική. Και για τα δύο σώματα. Αυτή είναι μια δυνατότητα. Ως προς τις δομές. Επίσης δυνατότητα υπάρχει και για διαρθρωτικούς δεσμούς. Κοινό καπέλο θα έλεγα μεταξύ των μελών της Eurogest και των Ευρωπαίων, των εθνικής προλεύσεως μελών της Eurogest και των εθνικών κατηγόρων συλλογική μορφή έχει προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται από τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Δεν θα υπάρχει ένας επικεφαλής κατήγορος. Συλλογικό όργανο, υπό το οποίο θα έχουμε αποσπασμένους κατηγόρους. Και άρα τα εθνικά μέρη της Eurochest μπορούν παράλληλα να υπηρετούν και ως Ευρωπαίοι κατήγοροι. λύση που έχουν υποστηρίξει τα μικρότερα κράτη. Άλλα κράτη όμως επικρίνουν αυτή τη δυνατότητα και τη λύση. Γιατί λένε θα οδηγούσε σε διπλές ε, αρμοδιότητες, αλλά με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Άρα συνεχίζει τη συζήτηση από ό,τι γνωρίζω στο θέμα αυτό. και στη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών υπάρχει το ζήτημα της υπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο σωμάτων. Προς το παρόν είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε περαιτέρω ανάλυση, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι δομικοί δεσμοί μεταξύ των δύο φορέων. Αλλά ασφαλώς θα χρειαστεί οπωσδήποτε συνεργασία και κυρίως ανταλλαγή πληροφοριών. Και εδώ έχουμε διάφορα σενάρια, όπως το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων της Eurojust, όπου θα μπορούσε το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων να είναι κοινό. Πρώτη δυνατότητα. Άλλη δυνατότητα, αμοιβαία προσφορά πρόσβασης στα δύο συστήματα διαχείρισης υποθέσεων με τη βάση του συστήματος hit no hit, με την αγαντανάκλαση της πληροφορίας δηλαδή, πρόσβαση στο περιεχόμενα του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. Much. I Τρεις ακόμα έχουν ζητήσει τον λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Βόνι από το ΕΛΚΑ. Πρώτα. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχω ερώτηση. Έχω όμως ανησυχία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εισηγήσεις σας. Πάρα πολύ χρήσιμες. Στην άλλη πλευρά όμως δείχνουν την έλλειψη συνεργασίας, την έλλειψη συνέπειας και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις και τις συστάσεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι αν, όπως ελπίζω, ε, θα έχουμε συνεργασία με το Συμβούλιο για τον Κανονισμό περί προστασίας ε, δεδομένων θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι που θα μοιάζει με εφαρμοστικό πακέτο και εκεί θα πρέπει να ε, βλέπουμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. θα πρέπει επίσης να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε αυτόν τον κανονισμό με τους κανόνες και με τις δραστηριότητες όλων αυτών των ευρωπαϊκών οργανισμών. Πιστεύω πως ε, ο ρόλος ε, του Ευρωπαίου κατηγόρου επόπτη δεδομένων είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον και γι' αυτό και θα πρέπει να έχει στη διάθεση του κάποια εργαλεία. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο μας ε, και να έχουμε δηλαδή κανονισμό και εφαρμοστικό πακέτο, θα πρέπει να αρχίσουμε τη δουλειά μας τώρα. Και η ανάλυση σας και τα διάφορα σενάρια που μας παρουσιάσατε είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρήσιμα Σας ευχαριστώ για την ε, εισήγηση που κάνατε, αλλά πρόκειται και για μια έκκληση για ευρύτερη συνεργασία στην Επιτροπή μας και στα θεσμικά όργανα. Διότι ε, χωρίς... Ε, μάλλον η έκθεση σας δείχνει ότι χωρίς ένα εφαρμοστικό πακέτο και πολύ πιο ε, ολοκληρωμένη λειτουργία όλων αυτών των ε, οργανισμών θα έχουμε πρόβλημα με την προστασία των δεδομένων και το σχετικό κανονισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρότασή μου είναι να ακούμε άμεσα τις απαντήσεις και εγώ ίσως να μπορούσα να προσθέσω τη δική μου ερώτηση σε αυτά που είπατε γιατί ακριβώς ε, αφορούσε το ίδιο πράγμα γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει οριζόντια ενοποιημένη προστασία δεδομένων και δεν ε, και τα, διάφορα σενάρια για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό ήταν ενδιαφέροντα. Απλά δεν υπήρξαν αρκετά προβλήματα, ε, μάλλον αρκετές προτάσεις όσον αφορά το προύμ ή τις βάσεις δεδομένων Όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στον προβληματισμό για τη ρύθμιση αυτού του πλαισίου. Πολλά θα χαθούν αν αφήσουμε Μάλλον, αναφερούσαμε τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων πρέπει να γίνεται διερκώς. Δεν είναι μία και μόνη λύση που ταιριάζει σε κάθε περίσταση και οι προστασίες, οι, προ, προκλήσεις μάλλον για την προστασία των δεδομένων σε σχέση με το ΣΕΝΚΕ δεν είναι οι ίδιες όσον αφορά το, το Europol. Η Europol ε, εξεργάζεται ε, πολύ ευαίσθητες πληροφορίες, ε, δικαιώματα πρόσβασης στους πολίτες και είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα εδώ. Γι' αυτό θα ήταν λάθος να σκεφτεί κανείς ότι Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα όργανο το οποίο όμως δεν θα δουλεύει. Κάθε φορά λοιπόν που δημιουργείται ένας οργανισμός, νέες εξουσίες δημιουργούνται και άρα πρέπει να περάσει ξανά η διαδικασία της προστασίας των δεδομένων από την ίδια διαδικασία. Γι' αυτό είμαι και υπέρ των κανόνων για την προστασία των δεδομένων που θα αντιποκρίνονται κάθε φορά στις συγκεκριμένε προκλήσεις όσον αφορά τις πολιτικές ελευθερίες. Όμως υπάρχουν πολλά στην προστασία των δεδομένων που μπορούν να διορθωθούν. Ε, και αυτό αφορά ίσως να αντιφάσκω, αλλά όχι κανονικά. Πάντως πρόκειται για το κεφάλαιο που αφορά τα δικαιώματα διόρθωσης ή πρόσβασης του ατόμου και το, το κεφάλαιο για την εξωτερική ανεξάρτητη εποπτεία. Και ε, πολύ είμαι ευχαριστημένο που ο βουλευτή Μπόνι υπογράμμισε ότι χρειάζεται ένα συνολικό πακέτο τώρα, διότι αν δεν έχουμε μια άποψη για την Κομισιόν για το τι θα, θα κάνουμε με τον επόπτη, είναι πρόβλημα. Ε, και βλέπω ότι η μεταρρύθμιση του Eurojust ε, φέρνει άλλες επιλογές διαφορετικές από αυτές στη Europol λόγω της αβεβαιότητας του τι θα γίνει με το EDPS. Και καταλαβαίνω απολύτως την αβεβαιότητα και τις αμφιβολίες και τους λόγους να προχωρήσει κανείς σε μια μεταρρύθμιση προς τη μια κατεύθυνση ενώ στην άλλη μεταρρύθμιση προς την άλλη κατεύθυνση. Όμως αυτές οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις δεν είναι ιδανικές. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε τους συγκεκριμένους κανόνες που να ταιριάζουν στους οργανισμούς και τις εξουσίες τους και αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα πακέτο για τις γενικές αρχές, τα γενικά δικαιώματα και την ιδέα της εποπτείας που θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών και επίσης στις ιδέες περί ορθής ε, χρηστής ε, ρύθμισης, κανονιστικής ρύθμισης. Γι' αυτό είναι αυτό το κομμάτι που λείπει τώρα από αυτό το puzzle, δηλαδή τι κάνουμε με τον επόπτη. Θα έπρεπε τώρα να το γνωρίζουμε πριν να μεταρρυθμιστεί το Eurojust και η Europol. Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε ότι τα όσα ακούσαμε στην πρώτη εισήγηση είναι ακόμα πιο σημαντικά αν Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων στι διάφορες ε, οργανισμούς, οπότε η, η ανταλλαγή πληροφοριών καθίσταται πιο περίπλοκη. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι δύο παρα, ε, παρουσιάσεις. Δεν υπάρχει νομίζω αντίφαση ως προς το να συνεργάζονται οι υπηρεσίες, η οικονομία δεδομένων, η υποχρέωση να κρατούνται κατά τρόπο ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα, ισχύει για κάθε τομέα, επομένως σε αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι χρειάζονται και συγκεκριμένε διατάξεις. και μια ανεξάρτητη αξιολόγηση, ουδέτερη αξιολόγηση, είναι επίσης πολύ σημαντική και μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε νέα δεδομένα. Αυτό είναι μια ε, αξιολόγηση η οποία πιστεύω ε, βρίσκει μεγάλη αποδοχή και απαντάται με πολύ ενθουσιασμό πολλούς. Στην ε, παρακολούθηση όμως της μεταφοράς δεδομένων θα ήθελα να σταθώ. Ένα θέμα το οποίο πάντοτε μας προσβληματίζει γιατί είναι διαφορετική η συστηματική. Άρα λοιπόν τεχνικά ποιος παρακολουθεί τη μεταφορά για να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλής, μεταφορά δεδομένων, και δεύτερον, για να περάσω και στην πρώτη παρατήρηση, ποιος παρακολουθεί, ποια είναι εκείνα τα δεδομένα που πάνε και σε ποιον πάνε τα συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των δύο υπηρεσιών όπως μας λέτε μεν, αλλά από την άλλη μας λέτε ότι το, η επιβολή του νόμου αφενός, ε, η δικαστική, ο δικαστικός χώρος αφετέρου έχουν διαφορετικά ε, καθήκοντα. Ποιος λοιπόν θα ελέγξει τι είδους δεδομένα περνάνε από τον ένα στον άλλον και πού τίθεται τα όρια στην τελευταία ανάλυση. Επίσης, για να το τραβήξω λίγο περισσότερο, ε, για τον Ευρωπαίο Δημόσιο Κατήγορο. Δεν θα κάνω ρωτήσει σχετικέ με τα προσωπικά δεδομένα, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει το θέμα, αν και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά με τη δομή που έχει αυτή τη στιγμή και προβλέπεται, έχουμε αφενός με τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, που δεν είναι και 100% ιδεώδης, έστω, λόγω και των ε, παραδόσεων των διαφορετικών, των αστυνομικών αρχών, των δικαστικών αρχών στα ε, κράτη-μέλη. Ποιος χρησιμοποιεί ποια υπηρεσία για ποια δουλειά και πού μπορεί να υπάρξει κάποια ε, δυσλειτουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά επίσης πρέπει να πούμε ότι και οι δημόσιοι κατήγοροι έχουν διαφορετικούς ρόλους με στα εθνικά κράτη. Αν λοιπόν σε αυτή την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας του Δημοσίου Κατηγόρου. Μπορούν και δουλέψουν πολύ διαφορετική προελεύσεως εθνική κατηγορία. Τι το ευρωπαϊκό μένει στον Ευρωπαίο Δημόσιο Κατήγορο, τι αρμοδιότητα του μένει, όχι μόνο σε σχέση με τη Europol, την Eurojust, αλλά και σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Πώς θα κρίνω εγώ μετά ποια δικαιώματα ή προνομίες έχει ο Εθνικός Δημόσιος Κατήγορος όταν ε, ο Ευρωπαϊκό Δημοσιοκατηγορό των Αθηνικό έχει τελείω διαφορετικέ αρμοδιότητε. Ή θα μπορεί να αποφασίζει, α, για να δω, να το ελέγξω αυτό, να κάνω μια, να ξεκινήσω μια δίωξη, ή δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ και θα πάω να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει πιστεύω να συστήσουμε εδώ, γενικότερα. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το περίπλοκο πλέγμα στα ευρωπαϊκά πράγματα και βέβαια με τη, με, τη διαφορά στις κατανομές και τους διαχωρισμούς σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των ε, υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε στις παρατηρήσεις αυτές. Θέλετε να προχωρήσουμε. Αν κατάλαβα όλα όσα μου είπατε και νομίζω τα κατάλαβα, λέει ο κύριος Δεχέρτ, συμφωνούμε απολύτως. Και προφανώς δεχόμεθα την αρχή της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών της αστυνομίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτονόητο και αλληλεξαρτώμενο είναι αυτά τα δύο. Θα πρέπει δηλαδή να δεχθεί και ο Πελίτη από πλευρά του ότι η, Πορτογαλία, η Πορτογαλική αστυνομία θα έχει την ίδια πρόσβαση στο φάκελό του με αυτήν που, έχει η, που έχουν οι οικίε αστυνομικέ αρχέ. Γιατί αυτό σημαίνει Ευρώπη στην τελευταία ανάλυση. Άρα θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δημοσίου Κατηγορού να έχει πολύ ισχυρό ρόλο και κεντρικό ρόλο. Το άλλο είναι ότι η Europol είχε ζητήματα σχετικά με την διαπραγμάτευση μεταφοράς δεδομένων ως προς, ή μάλλον προς χώρες που δεν έχουν επαρκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με τη Eurojust ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως εμείς πιστεύουμε ότι θέλουμε να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες, αλλά να μην έχουν τα παιχνιδάκια αυτά στα χέρια τους. Ή να υπάρχει μία ενιαία αλλά και στεναρή εποπτεία των δύο υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει και την συνοχή, γιατί αν δεν μπορεί μια υπηρεσία, μια χώρα να εξασφαλίσει εγγυήσει προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι αδύνατον να λειτουργήσει και δεν μπορεί μία να εγγυάται και άλλη να μην εγγυάται. Επομένως, ε, χρειάζεται κάποια εποπτεία και κάποια ισχυρή εντολή ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να περνάει από το κοινοβούλιο, κάθε εβδομάδα να περνάει από το κοινοβούλιο η υπόθεση αυτή της εποπτείας. Κύριε Βάιενμπεργκ, σε σχέση με την ερώτησή σας για τον έλεγχο των πληροφοριών, ξαναπερνάω στην αρχή του κατόχου, owner principle, σε σχέση με, τις, ε, με τη διάθεση των πληροφοριών. Οι εθνικές αρχές δηλαδή, αυτές που έχουν προσφέρει τις, τις ε, πληροφορίες, που έχουν διαθέσει πληροφορίες στην Europol, παραμένουν και κάτοχος της ε, πληροφορίας. Αυτό οδηγεί σε πολλά προβλήματα σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχει όμως και άλλο ζήτημα, όχι σχετικό. Ή μπορεί και να είναι. Ποιος ελέγχει την καλή ροή των πληροφοριών. Ποιος επαληθεύει την ε, αγαστή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και σωμάτων. Εδώ κάποιοι μηχανισμοί υπάρχουν με ένα είδος αξιολόγησης, ευρείας αξιολόγησης των σχέσεων μεταξύ των δύο υπηρεσιών και άλλων φορέων. Αλλά υπάρχει και μια, υπάρχει μια κάποια αδιαφάνεια ως προς την ε, έκβαση αυτής της αξιολόγησης. Ή αν κοιτάξουμε άλλους μηχανισμούς υφιστάμενους, τη σειρά των αμοιβαίων ε, συμφωνιών του 2010 μεταξύ Europol και Eurojust. Εκεί μια από τις τελικές διατάξεις αναφέρεται σε αξιολόγηση της ε, καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών και ότι θα πρέπει και οι δύο να λογοδοτούν ε, άπαξ το χρόνο στην Επιτροπή. Ωραία, αλλά γίνεται πραγματικά αξιολόγηση. Αυτό δεν το ξέρουμε. Άρα έχουμε και πρόβλημα διαφάνειας. Μια ιδέα, μια ιδέα βεβαίως θα ήταν να ε, προαγάγουμε αυτές τις ε, αξιολογήσεις αμοιβαίων σχέσεων, αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και των υπηρεσιών, μεταξύ υπηρεσιών και σωμάτων, με δυνατότητα εδώ να αναπτυχθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ίσως, ή θα μπορούσε να υπάρχει και ένας ε, ε, γύρος αμοιβαίων ε, αξιολογήσεων μεταξύ των υπηρεσιών για τις διυπηρεσιακές σχέσεις τους ακριβώς στον χώρο της ποινική δικαιοσύνης. Το άλλο θέμα που αναφέρατε ήταν το σχετικό με την προσθέμενη αξία. Βεβαίως και θα πρέπει να διακρίνουμε την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και το, την έκβαση των ε, τρέχουσων συνομιλιών. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η προσθέμενη αξία. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Και θα πάμε σε ενισχυμένη συνεργασία. Γιατί όσο υπάρχει η διαπραγμάτευση, τόσο προχωρούν και οι φιλοδοξίες. Τώρα φαίνεται να πηγαίνουν προς ένα κολυγιακό πρότυπο. Με, ερώτηση, με ερώτημα τι προσθεμένη αξία θα φέρουν σε σχέση με τη συλλογική δομή της Eurojust. Η απάντηση θα είναι ότι είναι διακυβερνητική η λογική συλλογική λογική της Eurojust, άρα μόνο υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει, ενώ ο κατήγορος, ακόμη και με συλλογική δομή, θα έχει να προσφέρει περισσότερα πράγματα. Θα είναι υπερεθνικός κατά βάση. Και άρα δεν θα είναι μόνο πάροχος υπηρεσιών. Αλλά θα έχει δεσμευτικέ εξουσίες επί των εθνικών αρχών. Συμφωνώ μας μαζί σας ότι όσο προχωρούν οι διαπραγματεύσει, τόσο και το ζήτημα της προσθεμένης αξίας προχωράει. Αλλά έχουμε ναι, εξέλιξη, EGN, κοινό δίκτυο, δικαστικό δίκτυο, Eurojust, με όχι τόσο καλές σχέσεις, μεταξύ τους και βέβαια εδώ θα πρέπει να δούμε ποια, κρίνεται πάντα ποια υπόθεση θα πάει στη Eurojust, ποια θα πάει στο δικαστικό δίκτυο και τώρα θα έχουμε και το δημόσιο κατήγορο. Ε, δεν θα είναι εύκολο για τον ε, ε, νομικό που ασχολείται με τέτοια θέματα να, να καταλάβει σε ποια υπηρεσία θα πάει μια υπόθεση. Και το εγχειρίδιο ακόμα που θα πρέπει να ορίσει ε, τις λεπτομέρειες θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ. Ίσως εδώ θα μπορούσαμε να ξαναδούμε το θέμα αυτό αύριο το πρωί που θα έχουμε τον πρόεδρο. Έτσι. Είναι θέμα διοργανικού συντονισμού. Αυτό είναι που επήγει. Ε, Μόνικα Χολμάιερ είναι η επόμενη που θέλει να ρωτήσει κάτι. Παρακαλώ. Όσο πιο πολλά ακούω, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνω ότι πρέπει να διευκρινιστεί η κατανομή και η συνεργασία μεταξύ ε, των διαφορών υπηρεσιών και τις υπηρεσίες ε, του Ευρωπαίου Κατηγόρου. Είναι πολύ επιφυλακτική και δυσπιστή εναντί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πολίτες. Η Eurojust κάνει δέκα των πόρων σε την Επιτροπή. Δεν μπορώ να πω ότι με πείθει το κατασκεύασμα αυτό και το αρχιτεκτόνιμο που βλέπω ότι οργανώνεται κατά ευρωπαϊκό τρόπο, κατά τρόπο αποτελεσματικό, όταν έχουμε οργανωμένο έγκλημα διεθνές, οργανωμένο ταχύτατα δρόν, δρούν ε, και που δεν περιμένει να λάβουμε εμεί αποφάσεις, ούτε λαμβάνει υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες του πνεύματος του θεσμικού που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν διερωτώ εάν ένα από τα ζητήματα που προκύπτει σε σχέση με την καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας είναι το εξής, ότι έχουμε μια πληθώρα δεδομένων, πληθώρα δεδομένων, αλλά ποιος είναι αυτός που εν τέλει θα τα πιάσει, θα τα ε, συγκεντρώσει, θα τα αναλύσει και θα δει, θα επιλέξει ποια είναι τα πιο σημαντικά. Και η μητέρα θα τα αξιοποιήσει, γιατί έχουμε τεράστιο όγκο δεδομένων. Έχω λοιπόν αυτό το προβληματισμό. Όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία κυκλοφορούν, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω είναι ορθά ή εσφαλμένα, γιατί δέχομαι ότι μπορεί να είναι πολλά από αυτά ορθά. Ερωτώ λοιπόν, θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει μια επαρκής ανάλυση, δυνατότητα μάλλον ανάλυσης και ε, στάθμισης σε επίπεδο των διαφόρων ε, φορέων. Και δεύτερον, η Όλαφ σε σχέση με τον Ευρωπαίο κατήγορο, τι σχέση έχει. Η Όλαφ θα έπρεπε ιδιαίτερα να λαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και ο δημόσιος κατήγορος θα έχει δημόσιες, θα έπρεπε να έχει διοκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες σε σχέση και με το οικονομικό έγκλημα. Όλαφ και ΕΠΟ λοιπόν, η δημόσιος κατήγορος, ε, δεν έχω δει ακριβώ πού διαχωρίζονται τα παιδιά αρμοδιοτήτων τους ή όπως είπατε νωρίτερα Eurojust και ΕΠΟ, Ευρωπαίος ε, κατήγορος. Ίσως θα είχε και νόημα να βάλουμε από, κάτω από την ίδια ομπρέλα τις τρεις υπηρεσίες και σιγά σιγά να οργανώσουμε την δομή τους ώστε αυτός ο αγώνας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος να μην γίνεται από το ένα θεσμικό όργανο, το ένα φορέα μέχρι τον άλλον, αλλά οργανωμένα και συντονισμένα. Για μην κάνει ο ένας το ένα πράγμα, ο άλλος να έχει δυνατότητα να κάνει μόνο το δεύτερο και ο τρίτος μόνο το κάτι άλλο. Γιατί είναι πολύ περίπλοκο όλο αυτό και, μέσα σε ένα... και μέχρι να τα εξηγήσουμε όλα αυτά έχει το οργανωμένο έγκλημα αναδιπλωθεί και ανα... Ε, αναπτυχθεί. Έχουμε πάρα πολύ, ε, πολλές δυνατότητες. Αν κοιτάξουμε την υπόθεση Φίλιπ Μόρις, όπου κερδίσαμε 10 δισεκατομμύρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή εργαστήκαμε καλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά το θέμα των δικαστικών μας δομών. Εδώ μια τεράστια ε, επιχείρηση, πολυεθνική επιχείρηση, η οποία συμμετέσχε και υποφελήθηκε από εγκληματικές δομές, πλουτίζοντας. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές από τέτοιες εγκληματικέ δραστηριότητες οι πιο μικροί, ένα πλοίο το οποίο συλλαμβάνεται στα νερά της Ελλάδας ας πούμε, ε, αντιμετωπίζουν τις συνέπειες, ε, τα πιο μικρά ψάρια του κυκλώματο αυτού, αλλά οι μεγάλοι, μεγάλες εταιρείε μπορούν να διαφεύγουν. Η Europol θα πρέπει βεβαίως να έχει τους εθνικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι πάγονται στην εθνική κυριαρχία, εκφράζουν τις εθνικές δομές και το καθεξής, αλλά ταυτόχρονα είναι μέλη ενεργά των ανακριτικών εργασιών που ε, αναπτύσσονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι απλό, αλλά και οι ανακριτικές δραστηριότητες που προχωρούν σε δικαστικό επίπεδο θα πρέπει να διευκρινιστούν γιατί είναι πολύ ασαφής ακόμα η εικόνα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Σχολιάστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας πρέπει να πω ότι συμφωνώ μαζί σας για το ότι χρειάζεται εξορθολογισμός. Και είναι αλήθεια, όταν αναφέρθηκα στους τρεις φορείς, πράγματι πρέπει και η Όλαφ να συμμετέχει μαζί με αυτούς τους τρεις. Και όταν μιλάμε για το μέλλον και για το πού θα εγκατασταθεί ο Ευρωπαίος εισαγγελέα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τα περιόλαφ. Θα εξακολουθεί να υπάρχει έτσι όπως έχει σήμερα, θα χωριστεί, θα περιοριστεί. Δεν νομίζω ότι είναι πια αμφιλεγόμενο το ότι πρέπει να μειωθεί όλαφ. Ακόμα και στα έγγραφα της Επιτροπής, κατά κάποιο τρόπο είναι σαφές ότι μέρος του προσωπικού της Όλαφ θα πρέπει να μεταφερθεί και να πάει στο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ξέρετε ότι μια από τις βασικές αρχές στην πρόταση της Επιτροπής ήταν να δημιουργήσει έναν Ευρωπαίο Εισαγγελέα με κόστος μηδέν. Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή μεταξύ άλλων, ήταν να μεταφέρει το προσωπικό της Όλαφ, η μέρος του, στο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Βέβαια, να υπάρξει τελικά αυτή η υπηρεσία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κόστος μηδέν ε, δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό. Αλλά αν μη τι άλλο, η προσπάθεια έτσι θα γίνει. Και η Eurojust εννοείται ότι ανησυχεί γιατί σκέφτονται κόστος μηδέν, μα θα λειτουργήσει καλά μετά. Η Eurojust, το γραφείο αυτό Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα από τα βασικά ερωτήματα βέβαια είναι το μέλλον τη Όλαφ πάντως. Είναι αλήθεια αυτό. Όταν μιλάμε για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Όλαφ μπαίνει βέβαια στο σκηνικό και αυτή. Τώρα για το άλλο θέμα, ναι. Αν κοιτάξουμε αυτή την αρχή του κόστους 0 και ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις διοικητικές διευκολύνσεις της Eurojust. Για να γίνει αυτό, εγώ δεν βλέπω δυνατότητα να εγκατασταθεί αλλού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρά μέσα στη Eurojust. Βέβαια το θέμα της έδρας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έχει λυθεί ακόμα. Το 2003 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέλαβε τη δέσμευση να εγκατασταθεί στο Λουξεμβούργο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά τώρα το θέμα είναι αν είναι στο Λουξεμβούργο, τότε πώς θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις διευκολύνσεις δωρεάν. Αν μείνουμε στην αρχή αυτή του κόστους μηδέν, που πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή, γιατί σημαίνει εξορθολογισμό, τότε θα πρέπει να εγκατασταθεί στη Χάγη. Τι θα γίνει όμως με την πολιτική δέσμευση που ανελήφθη απέναντι στο Λουξεμβούργο, ερωτηματικό. Πολλά είναι δηλαδή τα ζητήματα που μένουν να λυθούν και το θέμα της έδρας θα λυθεί στο τέλος της όλης διαδικασίας. Δεν θα ξέρουμε περισσότερα παρά πολύ αργότερα. Πρόεδρος, μην ξεχνάμε ότι τα θέματα έδρας είναι θέματα συμβουλίου. Έτσι. Και να θυμηθούμε επίσης ότι όσον αφορά αυτό τα θέματα ευρωπαϊκής διαδικασίας και Eurojust, οι διαδικασίες είναι διαφορετικές. Το ξέρουμε και εμείς αυτό. Πρέπει να λυθεί το διαδικαστικό πρώτα απ' όλα. Αν έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό, ευχαρίστω. Αλλά έχουμε κι άλλον έναν που θέλει να ρωτήσει κάτι. Η κυρία Λορεστίν, που είναι η συγγήτρια για την οδηγία όσον αφορά την προστασία δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου, Eurojust κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Λοριστίν, και ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές. Η εικόνα που παρουσιάζουν είναι θλιβερή όσον αφορά τις θεσμικές δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για 28 διαφορετικά συστήματα και νοτροπίες Τώρα πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε αυτό το 28 με 4, 5, 6 ή δεν ξέρω εγώ ποιον αριθμό. Ο δικός μας ο ρόλος εδώ είναι να δουλεύουμε πάνω σε οδηγίες και νομικά κείμενα, ελπίζοντας ότι κάποιος θα τα εφαρμόσει όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ένα μικρό κομματάκι των αλλαγών που μας περιμένουν. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο και την εφαρμογή. Γιατί μπορούμε να έχουμε στα χαρτιά ένα τέλειο σύστημα. Πώς θα λειτουργήσει όμως το σύστημα αυτό, πώς θα το εφαρμόσει ο κόσμος. Γι' αυτό και θέλω να αναφερθώ εδώ στην διαπαιδαγώγηση και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Κοιτά εδώ τους τίτλους σας. Ο καθηγητής Τεχέρτ είναι διευθυντή στο τμήμα διατομεακών νομικών σπουδών, βασικό μέλος της ομάδας ερευνών κλπ. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα της κατάρτισης στο δίκαιο γιατί παρεβαίνει παντού, είτε πρόκειται για αναλύσεις, είτε πρόκειται για τεχνολογία, είτε πρόκειται για κοινωνικές αναλύσεις. Είναι οριζόντιου χαρακτήρα το θέμα σας, οπότε εσείς τι λέτε, πώς μπορούμε στην Ευρώπη να έχουμε τους νομικούς, τους αστυνομικούς, τους πολιτικούς που θα ψηφίζουν νόμους που να μπορούν να προσανατολίζονται προς τις νέες δομές, να τις καταλαβαίνουν και να αντιλαμβάνονται πώς θα λειτουργούν όλα αυτά τα μέσα και από την άλλη μεριά τι θα κάνουμε με τους πολίτες. Γιατί πολύ ωραίες όλες αυτές οι ιδέες που συζητάμε. Έχουμε πολίτες που μπορούν να συμμετέχουν να συμφωνούν ή να διαφωνούν με κάτι ανάλογα με τους κινδύνους λοιπά. Αλλά τι γίνεται με τους υπόλοιπους και τι γίνεται με την οτροπία προστασίας δεδομένων που θα επηρεάσει την εφαρμογή των νόμων αυτών. Η νοοτροπία διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αλλιώς είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλιώς είναι στη Γερμανία. Ε, χώρες που είχαν ολοκληρωτικό παρελθόν οι πολίτες έχουν εντελώ διαφορετική νοοτροπία όσον αφορά τον ιδιωτικό βίο, την προστασία των δεδομένων, τη χρήση των τεχνολογιών και τους κινδύνους που ελοχεύει. Συνεπώς, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τη δουλειά μας όσον αφορά τις θεσμικές αλλαγές με τη δουλειά που κάνουμε όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων, των αξιωματούχων αλλά και των πολιτών Μπορούν αυτά να πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ και στρέφομαι προς εσάς για να το σχολιάσετε αυτό. Πάρα πολύ ε, ε, ευαίσθητη το ερώτημα που θέσατε. Με ρωτήσατε, εγώ είμαι γενικά αισιόδοξο άνθρωπος. Νομίζω ότι με το άρθρο 16 η Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, το δικαίωμα να σκεφτεί ε, εις βάθος το, προστασία των δεδομένων γιατί προβλέπει το άρθρο 90 για το, η νομοθεσία περί μη διακρίσεων μια ευρύτερη προσέγγιση δηλαδή ε, και όχι τόσο περιορισμένη όσον αφορά τα θέματα, τα διασυνοριακά και τα θέματα της ενέας αγοράς. Εγώ θεωρώ πως το άρθρο 16 είναι μια ανοιχτή, ένα κλειδί μάλλον για ανοιχτό προβληματισμό και ως εντολή για να σκεφτούμε πραγματικά τι θέλουμε να κάνουμε όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Η εποπτεία λοιπόν και η εξέταση των όσων έχουν γίνει στο παρελθόν ε, μας οδηγεί να, έχουμε, να είμαστε αισιόδοξοι. Και όσον αφορά αυτή τη διαδικασία μάθησης, έχει συμβεί και γίνονται βέβαια συναισθηματικές συζητήσεις σχετικά με τους εθνικούς δημόσιους κατηγόρους, σχετικά με τη μία θηρίδα κτλ. Αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία ευρωποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχουν φάσεις όπου αυτές οι, αυτά τα συναισθήματα ε, προκύπτουν και μας επιτρέπουν να ασκούμε και αυτοκριτική. Αν ευρωπαϊκές απαντήσεις δεν λειτουργούν, τότε θα πρέπει να επανέλθουμε στο σημείο εκκίνησης. Εάν η εγκύτητα σημαίνει ότι ένας Ισπανός θα πρέπει να μπορεί να πάει στον Ισπανό επόπτη και όχι στον Ιρλανδό, και αν αποδειχτεί πως ο Ιρλανδός ε, επόπτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους Ισπανούς πολίτες, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό το πολύ ισχυρό, τις πολύ ισχυρές ευρωπαϊκές αξίες τις οποίες εφαρμόζουμε σε σχέση με τις διαδικασίες ε, επεξεργασίας δεδομένων γιατί είναι μια διαδικασία που αναπόφευκτα δεν μπορούν όλοι να είναι 100% βέβαια για το τι θα λειτουργήσει ανα πάσα στιγμή, εγώ θεωρώ πως η συζήτηση που γίνεται σχετικά γίνεται με επικοδομητικό τρόπο και βλέπω ε, να γίνονται δύο βήματα μπρος, ένα πίσω και ούτω καθεξής. Με εντυπωσιάζει δηλαδή αυτή η διαδικασία και νομίζω πως αν όλα τα θέματα δουν τον κανόνα, τον, μάλλον τον νομοθεσία περί περιβάλλοντος ή περί των δεδομένων. Ε, πρόκειται για παραδείγματα που η Ευρώπη έχει δώσει, έχει προσφέρει, έχει δώσει προστεθέμενη αξία ε, και όπου ε, φαίνεται να έχει να δώσει περισσότερα και θα πρέπει να περιμένουμε. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι υπέρ της απόλυτης ελευθερίας ή της αυτοδιάθεσης. Εγώ δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα Ακόμα και αν τα διάφορα περιστατικά ερμηνεύονται διαφορετικά, οικοδόμηση δηλαδή μια ρεαλιστική ε, κουλτούρας περί δομένων υπάρχει, γίνεται. Επερώτηση. Εγώ συμμερίζομαι τον, την αισιοδοξία κάθε είδους, ε, αλλά το θέμα δεν είναι σχετικά με την... Ε, ε, διαδικασίες και τις διαβουλεύσεις. Ε, το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να οικοδομήσει το, τη σταδιοδρομία του. Στην, ε, εδώ εμείς φτιάχνουμε τέτοια, τέτοια ύλη στα πανεπιστήμια, αλλά για τη χώρα μου, την Εστονία που είναι στο προσκήνιο όσον αφορά την ε, ε, ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν ε, πολύ μικρά πολύ μικρή λίγη ύλη, λιγοστή ύλη για την προστασία των δεδομένων. Ενώ είναι δικηγόρος. Πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ύλη στα πανεπιστήμια. Να πούμε ότι υπάρχουν αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, επί του οποίου μπορούμε να βασιστούμε. Είναι επίγον το θέμα, δεν είναι δηλαδή μόνο μια μακρά διαδικασία μακροπρόθεσμη. Είναι, είναι και μακροπρόθεσμη, αλλά είναι και τεράστιο το θέμα και ίσως να σας ρωτήσω κι εγώ ε, τι έχετε εσείς να πείτε για το θέμα το εκπαιδευτικό και το θέμα της ε, ύλη. Είναι λεπτό το ζήτημα γιατί ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να παίξει ρόλο όσον αφορά την πιστοποίηση προσόντων κτλ. Ε, πτυχίων κτλ. Αλλά είναι όντω σημαντικό το θέμα. Ε, είμαι βέβαιος ότι υπάρχει επαγγελματισμό στον τομέα, υπάρχουν πολλές επασχόληση, υπάρχουν 28 επόπτες, πολλές ευκαιρίες για επασχόληση, 400 γραφεία προστασίας δεδομένων, χρειάζονται εκεί κόσμο. για πιστώνω και αυτό έχει, ε, ήταν μια από τις χαρές της ζωής μου, ότι εγώ ήμουν ένας μυστήριος τύπος που έκανε κάτι πολύ παράξενο πριν από 20 χρόνια και τώρα όλοι έρχονται σήμερα και με ρωτάνε τι είναι προστασία δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ήταν μόνο ανταγωνισμός και τώρα βλέπουμε ότι οι ε, δικηγόροι του ανταγωνισμού που κυριαρχούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για πολλά χρόνια αρχίζουν να σιωπούν, ενώ το θέμα της προστασίας δεδομένων αυτά μεγαλύτερη σημασία. Μένω λοιπόν αισιόδοξο το μήνυμα της προστασίας των δεδομένων δεν είναι απλά κάτι το περίεργο και το παράξενο. Εξαπλώνεται και στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Πολλά μπορεί να μάθει κανείς για την προστασία δεδομένων από τις πρώην από τις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ψηφιακό χάσμα ή τίποτα τέτοιο, αλλά βλέπω όλα είναι και περισσότερο πανεπιστήμια που ενσωματώνουν ε, στη διάφορα θέματα τους και ε, τα θέματα της προστασίας των δεδομένων. Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, τελειώνοντας, ότι απόψε συζητήσαμε ε, χρηματοπιστωτικά προγράμματα ε, στον τομέα της δικαιοσύνης για το θέμα και ίσως θα έχει νόημα να εξετάσουμε και να στηρίξουμε προγράμματα που στόχο έχουν να αναπτύξει η προστασία των δεδομένων, δηλαδή εκπαίδευση των νομικών. Θα πρέπει ίσως και αυτό κάπως να το εξετάσουμε. Εγώ στο τέλος θα ήθελα να ρωτήσω δύο ακόμα ερωτήσεις. Μπορείτε να μου απαντήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι. Η πρώτη είναι για, τον ε, καθηγητή, ε, για την καθηγητρία Βάιντεμπεργκ. Έχουμε στρατηγική ασφαλεία στην Ένωση. Ε, χρειάζεται επιβολή, μάλλον στρατηγική επιβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας επίσης. Ναι, ήταν η απάντηση μάλιστα. Και η επόμενη για τον Πολτεβέρτ. Μιλούσατε για το άρθρο 16 της συνθήκης της και ανεξάρτητη εποπτεία εγγεγραμμένη στη συνθήκη. Αν σας απευθυνόταν λοιπόν με ερώτηση, θα λέγατε ότι ε, καλύπτεται η τωρινή δομή της Europol και Eurojust. Απάντηση ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολύ δουλειά έχουμε στους τομείς που μας παρουσιάσατε. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας, για τις μελέτες σας. Ξέρω ότι ήταν μεγάλο κόπος. Τελικέ μελέτε θα έχουμε στο τέλος του χρόνου. Περιμένουμε με μεγάλη ευμονία να σα ξαναδούμε. Σα ευχαριστώ. Πρώτη φορά προεδρεύω. Ελπίζω να πήγαν όλα καλά. Όχι, δεν ήθελα και να με χειροκροτήσετε, λέγοντά το. Αλλά να, επί τη ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω του διερμηνεί, στου οποίου αξίζουν τα χειροκροτήματα. Κάνουν πολύ καλή δουλειά και ευχαριστούν πολύ επίση.